Eh, eh, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε την κυρία Ντέι παρούσα σήμερα. Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και όπως γνωρίζετε ένα από τα σημαντικά ζητήματα κατά την εξέταση της απαλλαγής για την Επιτροπή είναι οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που έχουμε αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητής λοιπόν θα λάβει το λόγο για να προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης. Θα δώσουμε το λόγο μετά στην κυρία Ντέη και σε όποιον άλλον το επιθυμεί από τους συναδέλφους μας. Και παρακαλώ τον κύριο Χατζημαρκάκη να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ίσως είναι καλύτερα εάν μιλήσω στα αγγλικά για λόγους επικοινωνία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είστε παρόντες. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ακροάσεις της Επιτροπής μας κατά τη διαδικασία της απαλλαγή. Θα ήθελα να αναφερθώ στην υποχρέωση για λογοδοσία με ευθύνη. Υποχρέωση για λογοδοσία με ευθύνη. Ολόκληρο το πλέγμα του συστήματος λογοδοσίας δείχνει ότι υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας και εκτελείται. Πολλά πράγματα προσφέρονται, πληροφορίες, υλικό για ανάγνωση. Το ερώτημα όμως είναι αν οι πληροφορίες που διατίθενται είναι και οι σωστές. Και μήπως τελικά ε, τα πολλά λόγια και τα πολλά στοιχεία είναι ένα προπέτασμα μόνο πίσω από το οποίο κρυβόμαστε για να αποκρύψουμε την απουσία ευθύνης, την ανευθυνότητα. Και υπογραμμίζω το εξή, ότι σε προηγούμενε ακροάσει, ιδιαίτερα με τον Επίτροπο Τσόλο, τον οποίο θέλω να κατονομάσω συγκεκριμένα, διότι έκανε εξαιρετικά καλή παρουσία εδώ. Είδαμε λοιπόν από τι τελευταίε ακροάσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει πολύ σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Πολύ σημαντική βελτίωση. Αυτό βέβαια και βάσει και χάρη στι προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε βέβαια την υπόθεση του κτηματολογίου στην Ελλάδα, όπου η Επιτροπή συνέχισε να καταβάλει τα ποσά και το κοινοβούλιο ύστερα από πολλά χρόνια, περίπου 10, άσκησε τελικά το δικαίωμα της κυρίας και επέτυχε το επιδιωκόμενο αποτελέσμα. Επομένως ήταν οι προσπάθειες μας, οι κοινέ προσπάθειες ναι, αλλά και οι πιέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις οποίες οφείλεται το αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε καταλήξει σήμερα. Βέβαια υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Και το κυριότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή σε επιμέρους επιτρόπους ή γενικούς ε, διευθυντές, αλλά υποχρεωτικά τη δίνουμε την απαλλαγή σε όλους μαζί. Άρα εσείς έχετε ευθύνη α, εκ των συνθήκων και για την νομιμότητα της καταβολής των ποσών. Εδώ λοιπόν υπάρχει το, ο, ο λάκκος στη φάβα αν θέλετε, ότι δηλαδή έχουμε μόνο μία σφαίρα και στρέφεται αυτή προς όλους σας και όλοι μαζί εσείς φέρετε συλλογικά την ευθύνη της ε, απόδοσης λογαριασμών. Πώς λοιπόν μπορούμε να γυρίσουμε το μήλο του περιστρόφου και να ξέρουμε πού θα στραφούμε, όταν ξέρουμε πού βρίσκονται τα κενά, πού βρίσκονται τα παραθυράκια, πρέπει και να τα ασφαλίσουμε και είναι πλέον πιστεύω η στιγμή να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα για ένα πολύ απλό λόγο. Η Επιτροπή στην τέλος των καθηκόντων τους δεν έχουν ιδιαίτερη ε, υπαγωγή ή δέσμευση στα όσα έχουν συμβεί πριν από 10-16 χρόνια. Ας ε, γυρίσουμε λοιπόν τον τροχό, μια και έχουμε νέους τώρα επιτρόπους. Αλλά ας δούμε ποια είναι τα παραθυράκια. Έχουμε σαφή παραθυράκια, έχουμε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που παρουσιάζει κενά και πρέπει να τα ασφαλίσουμε. Και έτσι λοιπόν, κυρία Γενική Γραμματεύ, έχουμε καταρχάς το ζήτημα των, του χάσματος μεταξύ Γενικών Διευθυντών και Επιτρόπων και το δεύτερο μεταξύ, γενικό, ε, μεταξύ Επιτρόπων και κρατών μελών, του εθνικού επέδου δηλαδή. Για όποιον δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό, αυτά τα δύο χάσματα, αυτά τα δύο κενά, η απουσία ε, λογοδοσίας τα τελευταία 16 χρόνια έχει οδηγήσει σε αρνητική βεβαίωση αξιοπιστίας από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου. Ας αναφερθώ λοιπόν τώρα στους γενικούς διευθυντές καταρχάς και το συλλογικό όργανο της Επιτροπής. Έχουμε υπόψη ε, την ε, διοικητική μεταρρύθμιση ε, με την, Επιτροπή Σαντέρ. Έχουμε βεβαίως υπόψη ότι θέλετε να καταστεί πιο υπεύθυνο το προσωπικό σας συνολικά και καταγράφουμε, βλέπουμε μάλλον πώς καταγράφεται αυτό στην εκτίσια έκθεση δραστηριοτήτων. Αυτές οι αιτήσει εκθέσεις δραστηριοτήτων, μας λέει η Επιτροπή, είναι οι πυλώνες της αρχιτεκτονικής, του πλέγματος δηλαδή ευθύνης και ανάθεση ευθυνών. Μέσα από αυτές εκφράζεται η ανάληψη ευθυνών σε επίπεδο επιτροπής. Ε, είμαι λοιπόν καταρχάς πολύ περίεργος να δω πώς θα χειριστείτε τη νέα έκθεση που αναμένεται το 2011 που είναι η έκθεση αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 318 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ συγκεκριμένα θέλω να δω όχι μόνο πως τα ζητήματα της ε, νόμιμότητας, της, συνόμη, της σύνομης δηλαδή λειτουργίας, αλλά και την επίτευξη των στόχων. Πώς θα επιτυχείτε τους στόχους σας. Ξέρω ότι δουλεύετε σκληρά πάνω σε αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό ε, και, και δύσκολο το πρόβλημα. Κάτι άλλο τώρα, οι εκθέσει δραστηριοτήτων από τι γενικέ σα ουσιαστικά αποτελούν μια δική σας εκδοχή της ιστορίας. Καταγράφουν μια δική σας εκδοχή της ε, ιστορίας. Μάλιστα το ελεκτικό συνέδριο της ε, καταγράφει ως ε, απογραφές ε, διαχείρισης και δηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη και αντικειμενική έπεψη που θα τη συνοδεύει. Πράγμα όμως το οποίο δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή εξωτερική αντικειμενική θεώρηση. Οι εσωτερικοί δημοσιονομικοί ελεγκτέ τη Γενική σα Διεύθυνση είναι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν στο δημοσιονομικό έλεγχο. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, ο κ. Γκρέπ, τον έχετε εδώ παρόν, ε, δεν έχει πραγματικό έλεγχο στη λειτουργία τη γενική Διεύθυνση. απλώ εποπτεύει, παρακολουθεί το κατά πόσον οι εσωτερικοί ελεγκτέ κάνουν καλά δουλειά του. Η έκθεση λοιπόν, οι εκθέσεις ε, της εκθέσεις δραστηριότητας των γενικών διευθυντών δεν επικυρώνονται από την Επιτροπή ως λογικό όργανο ούτε από τους επιμέρους επιτρόπους και δεν δηλώνεται τυπικά ότι έχει γίνει η σύνομη λειτουργία και η εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση τους κανονισμούς. Αυτά όσον αφορά την πολιτική ευθύνη. Η έκθεση συνθέσεως που συντάσσεται υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέως, υπό τη δική σας ευθύνη δηλαδή, ελέγχει την πληρότητα, αντικειμενικότητα, ορθότητα και την ευστοχία των δηλώσεων μας στις αιτήσει εκθέσεις λειτουργίας ή δραστηριοτήτων. Δηλαδή αποτελεί μόνο μία σύνοψη, μία περίληψη αυτών και οι δικέ μου επικρίσει έχουν μια πολύ πρακτική συνέπεια για το Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο θεωρητικέ, δηλαδή. Ερώτω πώ εμεί, ω αρχή υπεύθυνη για την απαλλαγή και φαίνεται ότι είμαστε η μόνη αρχή υπεύθυνη για την απαλλαγή εν προκειμένου, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν τα στοιχεία για τα οποία μα ε, κάνετε λόγο στι ε, εκθέσει ε, δραστηριοτήτων προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή. Και παραλαμβάνω υπάρχουν πολλά στοιχεία αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι εύστοχα και ορθά. Και χωρί να θέλω να σα κουράσω, θα ήθελα να σα ε, δώσω κάποια στοιχεία από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τη Γενική Διεύθυνσης Περιφερειακή Πολιτική τη Ρέτζιο, την τελευταία της μόνο παράγραφο, προκειμένου να εξηγήσω τι παίρνουμε εμεί από τι υπηρεσίε σα ω εκθέσει για να καταλάβετε τι εννοώ. Διαβάζω λοιπόν. Καταρχάς, ε, αφού επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα που να προσβάλλει τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την υπογραφή την έχει η υπογραφή του κυρίου Άνερ, που ήταν και παρόν εδώ. Και λέει λοιπόν από 38 εκ των 79 προγραμμάτων που εξετάστηκαν, η ε, Γενικός δεν έχει θετική βεβαίωση για την ομότητα και σκοπιμότητα των υφισταμένων πράξεων και συναλλαγών. Για τις λοιπές έχουν καταγραφεί σε πρόωρο στάδιο ατέλειες ή ανεπάρκειες πριν από την πρώτη πληρωμή. Ερωτώ λοιπόν, πώς είναι δυνατόν εμείς ως αρχή αρμόδια για την απαλλαγή να αποδεχθούμε τέτοια δήλωση. Μας λέτε ξεκάθαρα ότι δεν ελέγχετε το τι γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Επιτροπή ε, Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρώτο στάδιο να πει Φερρυπίν, στις ελληνικές αρχές, ωραίο το σχέδιό σας, αλλά δεν δικαιούται χρηματοδότηση, δεν μας αρέσει. Η συνήθις πρακτική, ύστερα από ένα εξάμεινο, ένα χρόνο κτλ. Και, και σιγά σιγά βέβαια πιέζει ο χρόνος, Άρα έρχεται όλο και πιο κοντά το τέλο, ε, η προθεσμία δηλαδή τη λειτουργία του κανονισμού, θα έρχονταν οι Έλληνε να υποβάλουν ένα άλλο σχέδιο. Όχι πολύ καλύτερο, αλλά θα σα πίεζαν κιόλα, σα πιέζουν κιόλα. Και θα λένε, μα τα χρειαζόμαστε τα λεφτά. Και θα σα θέλουν και τον Υπουργό, θα σα πει και ο Υπουργό, θέλω κι εγώ τα λεφτά. Και θα έρθει στι Βρυξέλλε και θα σα λέει, τα χρειάζομαι τα λεφτά. Ε, χρειάζομαι, μπορεί να έχω 20 δισεκατομμύρια, έχω μόνο απορροφήσει τα 4, τα 16 τα οποία όμω έχω δικαίωμα, τα θέλω τώρα. Και θα πει τότε ο Επίτροπο σα, ο Γενικό Διευθυντή, δεν ξέρουμε τελικά τι θα τα κάνουν τα λεφτά αυτά οι Έλληνε. Και αυτή είναι η διατύπωση. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή η διατύπωση. Αλλά να πάρτε τα τα λεφτά. Και χρόνια μόνο μετά αντιλαμβανόμεθα ότι ούτε είχε δικαίωμα να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο αυτό, ούτε ήταν σωστό, ούτε προσέφερε προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Άρα δεν άξιζε τα χρήματα που του δώσατε. Και γιατί να, πώς θα το εξηγήσω αυτό στον Ευρωπαϊκό φορολογούμενο. Αυτέ είναι οι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που ανέχεται και αποδέχεται όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να, να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την πρακτική. Και σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, εγώ λέγω ξεκάθαρα ότι για να γίνει η μεγάλη αυτή αλλαγή θέλετε χρειάζεστε σύμμαχο. Δεν καταφέρατε να το κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Η πρώτη Επιτροπή Μπαρόσο ξέρουμε ότι υιοθέτησε μια δήλωση με στόχο να ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα. Δεν τα κατάφερε. Τώρα έχουμε τη δεύτερη επιτροπή Μπαρόσο και θέλουμε να σας προσφέρουμε το εξής. Βοήθεια, αρρωγή, συνδρομή δηλαδή την όθηση που χρειάζεστε προκειμένου σε θέση να πείτε, την ενθάρρυνση, αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πείτε στους, στις αρχές τις εθνικές, δεν μπορούμε να σας θέσουμε τα χρήματα, διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα με την αρχή, την αρμόδια για την απαλλαγή του προϋπολογισμού. Και δεν είναι πια μόνο θεωρητική και ακαδημαϊκή συζήτηση, αλλά ουσιαστική. Και όπως είπα, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ακριβείς πληροφορίες, να είμαστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι ορθές. Ερωτώ λοιπόν και πάλι, η εσωτερική αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικός πώς θα αλλάξει, πώς θα γίνονται επιτόπου διερευνήσεις χωρίς συστήματα ε, συναγερμού, δηλαδή χωρίς ο κύριος Γκρέι να προειδοποιεί τους συναδέλφους του ότι πρόκειται να κάνει έλεγχο στη δουλειά τους. Πώς θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Και επίσης οι επίτροποι που έρχονται εδώ σε ακροάσεις, βέβαια εντάξει εσείς εδώ σήμερα υφίσταται το ίδιο ψήσιμο, αλλά πάση περιπτώσει οι συνάδελφοι σα, γενικοί διευθυντέ και λοιποί δεν υφίστανται αυτή την ακρόαση. Ο επίτροπος έρχεται και βάζει το κεφάλι του στον τορβά με την ακρόαση. Εκείνος λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Και σας διαβεβαιώ ότι ο επίτροπο τον οποίο αφορούσε που ήταν αρμόδιος για την ε, παράγραφο στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα δεν ήταν ενήμερο. Μέχρι που του το ανέφερα εγώ δεν ήξερε υπόψη του αυτή την ε, παράγραφο, αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με πολιτική ευθύνη και με απόδοση ευθυνών. Και αυτό πρέπει να αλλάξει πλέον. Για το δεύτερο χάσμα ή κενό, και ήδη το συζητήσαμε σε έναν βαθμό, Πρόκειται για το χάσμα μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών. Δεδομένου ότι 80% του ευρωπαϊκού προπολογισμού ε, προχωρεί εκτέλεση από εθνικά φορείς, ε, εθνικά όργανα, ε, έλαβε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου του 2008 να υπογράφει όχι μόνο ο διαχειριστή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από εθνικής πλευράς. Θέλουμε δηλαδή και ο Υπουργός των Οικονομικών να φέτει την υπογραφή του σε αυτή τη σχετική έκθεση. Και εδώ δίπλα μου ο Γιάν Μούλντερ ήταν πέρυσι ο μεγάλος αγωνιστής και πρωτοπόρος αυτού του ιδεοδούς που πέτυχε τελικά να επιβάλλει. Και αν κοιτάξετε τις κάτω χώρες, για την οποία ο ίδιος βέβαια είναι πολύ καλός γνώστης, ε, βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα της τελικής δήλωση δουλεύει πολύ αποτελεσματικά. Να δούμε λοιπόν, ο κύριος Μιούλτερ κατάφερε ως Ολλανδός βουλευτής με πολύ σκληρή δουλειά να πείσει την πατρίδα του και αυτό αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική. Αυτή τη βέλτιστη πρακτική θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα και δεν πιστεύουμε ότι οι εθνικές δηλώσεις ε, βέβαια εκτέλεσης ε, πρόκειται να επιλύσουν όλα τα προβλήματα αλλά αποτελούν μια πρώτη ε, βαθμίδα, ένα πρώτο βήμα και μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο πάντως ευθύνης και για εθνικούς υπουργούς και για περιφερειακούς σε μερικές περιπτώσεις υπουργούς και πάντως να αποτελέσουν έναν τρόπο ε, εντοπισμού προβλημάτων, γιατί μερικές φορές τα προβλήματα φαίνονται αόρατα, φαίνεται να μην τα θέλει να τα βλέπει μια κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε με τον τρόπο αυτό να εντοπίζουμε αδυναμίες και προβλήματα σε προγράμματα σε επίπεδο κρατών μελών. Μήπως είναι τελικά γραφειοκρατική εφεύρεση. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι όχι, οπωσδήποτε όχι. Βεβαίως έχει τίμημα ε, η αρχή της ε, και της ε, απόδοση λογαριασμών. Αλλά πριν πούμε τι κοστίζει σε γραφειοκρατία, καλό θα είναι να δούμε και πόσο έχουμε χάσει, πόσο μας έχει κοστίσει η αναποτελεσματική διαχείριση, η κακή διαχείριση. Και στην παράγραφο 435 στην έκθεση του Ελεκτικό Συνέδριο, έκθεση του 2009, ετήσια έκθεση, αναφέρει ότι τουλάχιστον 30% των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο κρατών μελών πριν αυτή η δήλωση να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σας διαβεβαιώ όμω τελικά αυτό δεν έχει γίνει γιατί το φαινόμενο που περιέγραψα νωρίτερα με τον Έλληνα Υπουργό που έρχεται στις Βρυξέλλε και ζητάει τα λεφτά είναι καθημερινό φαινόμενο στις Βρυξέλλε. Και το 30% το έχουν ξεπεράσει τα πραγματικά στοιχεία νομίζουμε. Άρα η τρέχουσα διαχείριση, και, ε, μάλλον ο έλεγχος τρέχουσας διαχείρισης και λογαριασμών θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό και δεν, ε, δεν αρκούν αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής. Ξέρουμε ποια είναι η πάγια απάντηση της Επιτροπής μας. Λέτε δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα, ε, κάποιο σφάλμα που δεν εντοπίστηκε και δεν διορθώθηκε σε πρώιμο στάδιο θα ε, εντοπιστεί και θα διορθωθεί σε μεταγενέστερο. Αληθεύει όμως αυτό. Και να εδώ σε αυτούς τους λογαριασμούς που ευχαριστούμε πάρα πολύ που τους δημοσιεύσατε γιατί δημοσιεύεται όχι μόνο τις διορθώσεις στην ετήσια έκθεση λογαριασμών 4,8 δισεκατομμύρια είναι το ποσό των διορθώσεων, αλλά και τις ανακτήσεις 709 εκατομμύρια, το ένα δέκατο δηλαδή μόνο. Ευχαριστώ όμως επίσης και για τον ε, κατάλογο των ονομάτων. Είναι η πρώτη φορά που χωρίς απαραίτητα να θέλω να πω ότι ξεπροστιάζουμε κάποιους, πάντως ε, εξασφαλίστε κάποια διαφάνεια. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο θέλουμε να προαγάγουμε και στη τελευταία ανάλυση αυτό μας οφείλουν και τα κράτη-μέλη. Τους δίνουμε τα χρήματα, βλέπουμε ότι δεν γίνεται η χρήση τους σύνομα, μερικές φορές είναι και παράτυπη ε, η παράνομη χρήση τους και θα πρέπει να διορθωθούν αυτά. Το 1 δέκατο των 7,9 δισεκατομμυρίων είναι πολύ χαμηλό ποσοστό ανάκτησης κονδυλίων. Και πρέπει αυτό να προχωρήσει σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι μόνο μερικό αποτελεσματικό όπω επισημαίνει το Ελεκτικό συνέδριο και σημειώνω ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέλτιστη πρακτική σε επίπεδο επιτροπή αποτελεί ο τομέα τη γεωργία. Λειτουργεί πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, όχι σε, στον ίδιο βαθμό σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά το, ο συνολικό, ο μέσο όρο τη αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ καλό στη γεωργία. Στη συνοχή δεν έχουμε καλό ε, καλές επιδόσεις, 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα που βέβαια περιπλέκουν πολύ την κατάσταση και, θα πρέπει, και αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει επίσης να το ε, επικρίνουμε γιατί οι περίπλοκες διατάξεις και οι μηχανισμοί αποτελούν επίσης ένα άλλο προπέτασμα από το οποίο μπορεί κανείς να κρυφτεί αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορείτε να αναλάβετε δράση άμεσα. Ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν με τον Επίτροπο Άντορ υπεύθυνο για τα κοινωνικά ταμεία. Όταν ο επίτροπο Άντορ εντόπισε σφάλμα σε πρώιμο στάδιο, ξέρετε τι έκανε. Διέκοψε, δεν ήρε την ε, λειτουργία, αλλά διέκοψε αμέσως την καταβολή των ποσών. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο μέτρο, διότι ε, διδάσκει στα κράτη-μέλη ότι είναι υποχρεωμένα να τηρούν τους κανόνες αυστηρά. Και εγώ ε, τιμώ τον Επίτροπο Άντορ για την απόφαση αυτή και τη διακοπή, αλλά βέβαια ενδεχομένω και τη άλση, εφόσον χρειαστεί, δηλαδή εφόσον χρειαστεί ύστερα από εξάμεινο επανελειμμένων σφαλμάτων. Διαπιστώνουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη ότι υπάρχει σταθερή, μόνιμη ε, συμπεριφορά υποβολής κακών και μη δικαιούχων ουσιαστικά προγραμμάτων, ίσω γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο, γιατί ε, δεν, λειτουργούν οι υπηρεσίε σωστά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι που πρέπει εμεί να συζητήσουμε και στην Επιτροπή μα, βέβαια, ε, και στο πώ μπορεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένα ενδεχομένω κράτη-μέλη να παρεμβαίνει ε, απευθεία σε ορισμένα μόνο γιατί σε άλλα δεν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, αλλά σε ορισμένες εθνικές υπηρεσίες τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε ανοιχτά. Θα έλεγα λοιπόν επίσης να αναλογιστούμε και πάλι τις διάφορες αρχές Φερρυπίν την αρχή της ε, κοινή διαχείρισης, γιατί δεν σας απαλλάσσει των ευθυνών σας η ε, συνθήκη. Μπορεί να μιλάει για κοινή διαχείριση, αλλά τα 7,9 δις εσείς τα οφείλετε. Εσείς πρέπει να δώσετε λογαριασμό που βρίσκονται και πώς δαπανήθηκαν. Και εν τέλει, ο κύριος Λαμασούρ από την ε, Επιτροπή των Προϋπολογισμών, την αδελφή Επιτροπή, δεν είχε υπόψη τα ποσά αυτά, αλλά του τράβηξαν το ενδιαφέρον. Και γιατί, διότι Είχαμε διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου που αφορούσαν κονδύλια μη απορροφηθέντα και που είχαν μείνει στους λογαριασμούς μας στο τέλος του χρόνου και λέγαμε τι πρέπει να τα κάνουμε τα χρήματα αυτά. Ο κύριος Δαμασούρ λοιπόν είχε την εξή ιδέα να διασυνδεθούν αυτές οι μη υλοποιηθήσεις διορθώσεις, χρήματα δηλαδή τα οποία κακώς είχαν ε, χορηγηθεί και χρήματα τα οποία επιστρέφουν στους Υπουργούς των Οικονομικών. Και κυρία Ντέι, νομίζω ότι θα μπορούσαμε αυτή την ιδέα να την επεξεργαστούμε περισσότερο, να συνδέσουμε δηλαδή αυτές τις δύο κατηγορίες ποσών, γιατί νομικά δεν υπάρχει καμία ε, δέσμευση ω προ το αν τα χρήματα αυτά θα μένουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή αν θα επιστρέφουν στου εθνικού προπολογισμού. Με βάση συνθήκη τη Λισαβόνα δεν είναι σαφέ αυτό. Και άρα ο τρόπο με τον οποίο είτε θα κλείσουμε την υπόθεση είτε θα σφραγίσουμε τα χρήματα αυτά στους δικούς μας προϋπολογισμούς, στους δικούς μας λογαριασμούς, ίσως αποτελέσει και τον τρόπο να πιέσουμε τα κράτη-μέλη, να ξέρουν ότι τα χρήματα θα τα χάσουν εν τέλει. Αυτό πρέπει να το συστήσουμε και σε επίπεδο των Προϋπολογισμών. Και για να ολοκληρώνω, θα ρωτήσω εάν σκοπεύετε να αναλάβετε την πρωτοβουλία για διεξαγωγή μιας πλήρους αντικειμενικής και διεξοδικής αξιολόγησης της ε, ακρίβειας, ορθότητας και σκοπιμότητας των μηχανισμών που λειτουργούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη αρχιτεκτονική δηλαδή αυτής διαχείριση και ε, κατά τρόπον ε, ώστε να χορηγείται μια έκθεση δραστηριοτήτων ε, για την εκτέλεση των ε, σχετικών πράξεων και κονδυλίων ε, αξιόπιστη. Και εάν ο ιστορικό σα δημοσιονομική ελεγκτή, η επικεφαλή δημοσιονομική ελεγκτή, κύριο Γκρέι, θεωρείται ότι στη θέση που βρίσκεται και με δεδομένο το μηχανισμό δυνάμει του οποίου λειτουργεί μπορεί να επιτελέσει το έργο του αποτελεσματικά γιατί βέβαια τώρα έχει χορηγηθεί σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων η αρμοδιότητα για τον εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο και αν πρόκειται να κάνει απροειδοποιεί του εσωτερικούς δημοσιονομικούς ελέγχους ο κύριος Γκρέι από τη θέση που βρίσκεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχάς για τις γραπτές σας απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μας που μας καθοδηγούν στην έκθεση για την απαλλαγή, στις δραστηριότητες για την απαλλαγή. Σα ευχαριστώ για αυτέ λοιπόν και περιμένω βέβαια τι απαντήσει. σα. Ευχαριστώ. Uh, ε, ευχαριστώ, Γιώργο. Στην αρχή της συνεδρίασης έκανα ένα μικρό λάθος, ε, γιατί έχουμε εδώ και εκπροσωπό του ελεκτικού συνεδρίου. Αναφέραμε ότι θα είναι εδώ ο κύριος Γκαλέα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μεταβεί σε μία κηδεία στη Μάλτα, οπότε τον αντικαθιστά ο αδερφό του. Αν θέλετε λοιπόν, ε, κύριε Γενική Γραμματέα, να δώσω πρώτα το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο και μετά σε εσά. Ε, και θα ήθελα λίγο να ξέρω και ποιοι θέλουν να λάβουν το λόγο για να υπολογίσω και λίγο το χρόνο της συζήτησης. Ο κύριος Σουσί, λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ο συνάδελφος ε, Λουίς Γκαλέα, όπως είπατε σωστά κύριε Πρόεδρε, ε, κλήθη εχθές και πρέπει να πάει σε μια κηδεία στη Μάλτα. Να σας παρουσιάσω λοιπόν την έκθεση για το κεφάλαιο 9 του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για την ετήσια έκθεσή μας ε, για τα πεπραγμένα μέχρι τούδε. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης αξιολόγησης ε, ε, των δαπανών των ε, θεσμικών οργάνων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κεφάλαιο αυτό το, συνέδριο κάνει μια συνολική αξιολόγηση για τις δαπάνες για όλους τους φορείς και τα θεσμικά όργανα από κοινού βάσει ενός τυχαίου δείγματος συναλλαγών που αφορούν όλα τα όργανα. Ο απολογισμός είναι θετικός και το συνέδριο κατάφερε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πάνε στο 2009 ήταν νόμιμες και ε, νομότυπες. Ε, ε, αντίστοιχη κατάσταση είχαμε και το 2008. Κύριε Πρόεδρε, το ελεκτικό συνέδριο έκανε και κάποιες επιπλέον εργασίες. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να σας ε, θέσουμε και κάποιες παρατηρήσεις για καθένα από τα όργανα και φορείς. Ε, αφορά συγκεκριμένα θέματα. Πέρσι ασχολήθηκαμε ε, με την πρόσληψη ε, προσωρινά απασχολούμενων και ε, συμβάσεις οι οποίες προκύπτουν από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ε, με επίγον χαρακτήρα. Το συνέδριο κατέληξε στα εξή τρία σχόλια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, οι πρώτες δύο παρατηρήσεις αφορούν πληροφορίες οι οποίες διατίθενται στο Γραφείο Πληρωμών και στη Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ και εκεί ζητείται να γίνει σωστός υπολογισμός των επιδομάτων του προσωπικού διότι διαπιστώσαμε ότι δεν είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία και κάποια επιδέματα τα οποία καταβάλλονται μπορεί να μην είναι σωστά. Μία ακόμα παρατήρηση αφορά την αναθεώρηση ε, για τις ε, συντάξεις, ε, ε, διότι και εκεί διαπιστώσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και έγιναν και κάποιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες εκθέσεις και δύο σχόλια αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, αναφερθήκαμε στην, στους ανεπαρκείς ελέγχους πριν από την εφαρμογή του συστήματος ατομικών δικαιωμάτων, του ΙΡΙΣ, το οποίο είχε προβλήματα στον υπολογισμό των μισθών και ε, γι' αυτό και σταμάτησε η χρήση του Άιρες. Δεύτερον, είχαμε τους προσωρινούς κανόνες για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα για το τοπικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται στις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί ε, υπήρχαν προβλήματα για τα... Ε, δικαιώματα του προσωπικού και δεν λήφθησαν και κατάλληλα μέτρα για τη διευθέτησή τους εξετάστηκαν οι συνθήκες πρόληψης ε, των υπαλλήλων και ε, η δημιουργία του EAS. Αυτή ήταν μια σύνοψη των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε ερωτήσεις ε, και να ευχαριστήσω και εσάς και τους συναδέλφους σας για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ντέι για να ε, κάνετε μια πρώτη παρουσίαση και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ένα από τα βασικά ε, στοιχεία που ανέφερε ο εισηγητής ε, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιδιώκει να έχει μια επικοδομητική συνεργασία και διαπιστώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις πολλές από τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγώ είμαι η πρώτη που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά του ποιο είναι υπόλογο και ποιο έχει την ευθύνη για τα θέματα. Γνωρίζω τις πληροφορίες αυτές, γνωρίζω ότι είναι σωστές, θεωρώ μάλλον ότι είναι σωστές και νομίζω ότι εξαρτάται από το τι ψάχνει κάποιος. Ε, και αν υπάρχουν προβλήματα ε, πολλές φορές κάλλιστα μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αλλά η απάντηση είναι πάντα ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες. Το θέμα είναι πού θα τις βρούμε. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε καμία περίπτωση δεν ε, ε, είναι, δεν θεωρεί ότι έχει κάνει τα πάντα σωστά, αλλά είμαστε περήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει και αυτό αναγνωρίζεται και από τους εξωτερικούς μας ελεγκτές που είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Κάνει μια θετική αξιολόγηση των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρεί ότι βελτιώνεται η κατάσταση των σφαλμάτων και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή ε, βελτίωση σε αυτή την περίπτωση και τα πρόσφατα σχόλια, ε, χρόνια σχολίασαν και τις ε, ε διαχείριση ως προς το ποιος είναι υπόλογος και τι ευθύνες υπάρχουν όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Να σας αναφέρω τρία από τα βασικά θέματα. Το πρώτο αφορά το ποιος είναι, το υπόλογος και το ποιος έχει την ευθύνη. Η άποψή μου, επειδή βίωσε και το προηγούμενο ε, σύστημα και το τωρινό, ε, θεωρώ ότι είναι μακράν καλύτερο το νέο σύστημα και για τις δύο περιπτώσεις. Θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάναμε με τη μεταρρύθμιση είναι το γεγονός ότι η Γενική Διευθυντής είναι προσωπικά υπεύθυνη για την ε, διάθεση των πόρων που έχει κάθε τμήμα. Αυτό άλλαξε άρδιν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν χρήζει ακόμα βελτιώσεων, αλλά νομίζω ότι η πιο βασική αλλαγή έχει γίνει. Προσωπικώς δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ένα μείγμα των δύο συστημάτων. Ή θα έχετε ένα κεντρικό σύστημα το οποίο το επιλέξαμε και διαπιστώσαμε ότι δεν μας προστάτευε από τα σφάλματα και τις δυσκολίε. και επίση διαπιστώσαμε ότι ήταν μια πολύ μακροχρόνια και γραφειοκρατική διαδικασία και τελικώ αυτοί οι οποίοι λάμβαναν τι αποφάσει δεν είχαν την ευθύνη. Ε, ειλικρινά θεωρώ ότι το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όπου κάθε γενικό διευθυντή είναι υπεύθυνο, είναι καλύτερο, διότι μα δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε καλύτερα του πόρου που διαχειρίζεται ε, κάθε ε, πτυχή της πολιτικής και μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη ποιότητα συζήτησης μεταξύ Γενικού Διευθυντή και του Αρμόδιου Επιτρόπου και επίσης ε, η ευθύνη εναπόκειται εκεί που θα έπρεπε να εναπόκειται σε αυτούς που λαμβάνουν καθημερινώς τις αποφάσεις για την ε, διαχείριση της διεύθυνσης και θα έρθω κάποια στιγμή και στο θέμα της κοινή διαχείρισης ε, που είναι ένα διαφορετικό σύστημα προς συζήτηση. θεωρώ το σύστημα, ότι το σύστημα της αποκεντρωμένης ευθύνης είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική και σωστή διαχείριση. Το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για να ετοιμάσει την ε, έκθεση ε, πεπραγμένων δεν σημαίνει ότι κάνουμε απλώς μια σύνοψη. Ε, σε μια προηγούμενη μου επίσκεψη εξήγησα σε τι βαθμό ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προπολογισμών εργάζεται όλο το χρόνο σε όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές αλλά και για να βρίσκουμε και τους λόγους για τους οποίους εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις, εκθέσεις ή αποφασίζουν να μην παρουσιάσουν καμία επιφύλαξη και για κάθε επιφύλαξη που παρουσιάζεται φροντίζουμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα πρόγραμμα για την παρακολούθηση του θέματο. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν, υπάρχει διαφορετικό αριθμό επιφυλάξεων κάθε χρόνο και ε, δεν υπάρχει κάποια πολιτική που λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία επιφύλαξη. Εγώ ποτέ δεν θα παρέμβω στα όσα κάνει ένα γενικό διευθυντή για να του πω αν θα έχει ή δεν θα έχει επιφυλάξει. αλλά πάντα συζητώ μαζί του για ποιο λόγο θεωρεί ότι θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια επιφύλαξη. Και θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία συνεχού ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση. ε, παρά το γεγονό ότι ε, εξακολουθεί να δίνει την ευθύνη στο Γενικό Διευθυντή, μας έχει προσφέρει κάποιες βελτιώσεις. Έχουμε κάποιες πιο ε, στάνταρ αν θέλετε εκθέσεις. Έχουμε λάβει υπόψη και αυτά που μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο και το σχολίασε και θετικά το συνέδριο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει βελτίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και εξακολουθεί να διατηρεί το στρατηγικό στόχο του να ελέγχει τι κάνει και νομίζω ότι αυτό ε, αντικατοπτρίζεται θετικά και στο σύστημα. Δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχία το γεγονός ότι δεν το έχουμε επιτύχει ακόμα. Θεωρώ ότι είναι ε, μία ένδειξη ότι έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε και το χάσμα μειώνεται κάθε χρόνο. Επομένως είμαστε σε διαδικασία βελτίωσης. Τα όσα έχουμε τώρα έχει οδηγήσει και θα οδηγήσει σε συνεχή βελτίωση και νομίζω ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον μας να ε, αλλάξουμε το σύστημα εισαγάγοντα συστήματα για πιο κεντρική πολιτική ε, όταν έχουμε ένα σύστημα που φέρνει συνεχώς νέες βελτιώσεις. Τώρα, όσον αφορά τι αντιδράσει των κρατών μελών σε προτάσει που έγιναν εδώ στην Επιτροπή και έλαβε υπόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί είμαστε υπέρ των ε, εθνικών δηλώσεων, τι έχουμε δοκιμάσει, τι ε, έχουμε δει, ε, αλλά την απέρριψαν. Εσεί αναφερθήκατε στο περιορισμένο παράδειγμα ενός μικρού αριθμού κρατών μελών που ο καθένας ακολούθησε με διαφορετική άγουσα για να το χρησιμοποιήσει. Εμείς το υποστηρίζουμε, τους υποστηρίζουμε αλλά προς το παρόν να σας πω ότι τα επιχειρήματα που έχουμε παρουσιάσει δυστυχώς δεν έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Ω προ την επανεξέταση των συστημάτων, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε πάντα κατά νου. Φέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάποιε προτάσει για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ίσω θα έχετε διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίασε και μια αναθεώρηση πέρσι και σκοπεύουμε να κάνουμε πάρα πολλέ αλλαγέ για τα συστήματα ελέγχων σε γενικές γραμμές θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη απλούστευση ε, στη διαχείριση των κονδυλίων. Αυτό νομίζω ότι αποκρίνεται και σε πολύ πιεστικές αιτήσει ε, των όσων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε και την υποστήριξη των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου για να ε, στοχεύουμε ακριβώς την απλούστευση όταν θα παρουσιάζουμε στις προτάσεις μας. Δεύτερον, ως προς τη συνοχή, θέλουμε να αυξήσουμε πολύ σημαντικά το βαθμό ευθύνη των κρατών μελών. Θέλουμε να απομακρυνθούμε από αυτή την ε, πολιτική του ο καθένα έχει δικαίωμα σε κάτι και ιδίω για τα διαστατικά ε, ταμεία να πούμε ότι τα κονδύλια δίνονται για να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Προ το παρόν λοιπόν εξετάζουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια μορφή σύμβαση με τα κράτη-μέλη όπου θα έχουμε εκ των προτέρων καταγεγραμμένα τα αποτελέσματα που περιμένουμε ώστε να έχουμε και την ανάλογη χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη. Αυτό φυσικά θα διαφέρει ένα κράτος μέλος, όχι μόνο λόγω του διαφορετικού συστήματος διακυβέρνηση, αλλά και λόγω του διαφορετικού βαθμού διοικητικών δυνατοτήτων. Ε, εσείς ε, υπονοείτε κάποια πράγματα, αλλά εμείς ε, θέλουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διοικητικές τους δυνατότητες, ίσως όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, για να τους παρέχουμε οικονομική συνδρομή αλλά και υποστήριξη. Και για να μην μακρηγορήσω άλλο, ε, θέσετε και μια πολύ ευθεία ερώτηση προς εμένα για το κατά πόσο θεωρώ ότι ο εσωτερικό ελεγκτή μπόρεσε να διεξάγει σωστά τα καθήκοντά του. Σα απαντώ λοιπόν σαφώ ναι. Έχει κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δυνατότητε εσωτερικών ελέγχων ε, είναι απευθεία ε, ε, δυνατότητε του Γενικού Διευθυντή και όλε οι εκθέσει πηγαίνουν στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και φυσικά στο ελεγκτικό συνέδριο. Θεωρώ λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της ποιότητας ε, της λειτουργίας της αρχιτεκτονικής δομής Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου και επιπλέον η κάθε μία από τις δομές που έχουμε εμεί ε, για εσωτερικό έλεγχο υπόκειται και μια ε, αξιολόγηση ποιότητας. Επομένως το όλο σύστημα είναι στημένο έτσι ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τον κώρικα δεοντολογίας και τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να τηρούνται. Ε, κάθε χρόνο έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν επαναπαυόμαστε όπως σας είπα. Προσπαθούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα αλλά έχουμε και ένα σύστημα το οποίο υπόκειται και σε εξωτερικό έλεγχο και παλήθευση και έχει περάσει και διεθνώς αναγνωρισμένους ελέγχους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω αργότερα αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ κύριος Χατζημαρκάκης. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσει λίγο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλερ. Ναι, ευχαριστώ. Με χαρά πάντα. Βλέπουμε την Επιτροπή, στην Επιτροπή μας την ε, κυρία Γενική Γραμματέα. Επιτρέψτε όμως κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα προς το παρόν. Ε, ασχολούμαι διεξοδικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διοικητικό όργανο, διοικητική αρχή και ε, διαρωτώμεθα εάν λειτουργεί όπως πρέπει Ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Ασχολούμαι λοιπόν, όπω είπαμε, την Επιτροπή και τον κανονισμό προσωπικού και ιδιαίω την απουσία από το χώρο, χώρο εργασία. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αρκετά γενναιόδορη ρύθμιση, όταν δηλαδή έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες ε, του κανονισμού, και μπορεί να αποσιάζει ένας ε, υπάλληλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι 12 έως 14 εβδομάδες από το χώρο εργασίας του. Πολύ γενναιόδωρο αυτό. Πράγμα το οποίο έχει για το 2009 συνολικά ε, κοστίσει 100.000 ημέρες εργασίας. 35 δηλαδή πλήρης θέσεις εργασίας. και ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε με θέσεις που δεν ξέρουμε ε, ποιος μπορεί να τι εγκαταστήσει. Έχουμε να κάνουμε με θέσεις που είναι αδρά αμοιβόμενε μερικές φορές, γενικού διευθυντέ. φερρυπίν. Και αν διαπιστώσουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μεγάλη, μεγάλο ποσοστό απουσίας, απουσίες ε, επί παραδείγματι σε ημέρες που δεν υπάρχουν ε, ούτε άδειες, ούτε αργίες, ούτε τίποτα, ούτε θρησκευτικές, ούτε εθνικές αργίες και βλέπουμε ότι ο Γενικός Διευθυντής έχει απουσία 9 ημερών αδικαιολόγητη, χωρίς να πάρει άδεια, την οποία υποχρεούται να πάρει κάποιος άλλος υπάλληλος σε κάποια άλλη υπηρεσία, τότε έχουμε να πούμε ότι μας κοστίζει το ισοδύναμο 150 με 180 θέσεις εργασίας ένας Γενικός Διευθυντής για την απουσία του αυτή στον χρόνο. Είναι πολύ γενναιόδωρος λοιπόν αυτός ο κανονισμός για τις απουσίες. Πώς θα το ρυθμίσει αυτό η Επιτροπή. Ναι, βλέπουμε στην απάντησή της ε, Επιτροπής ότι όλα είναι καλά, όλα τα έχουμε ρυθμίσει κατά τρόπο εύστοχο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα τροποποιήσουμε. Είναι δυνατόν όμως να έχουμε ε, ελεύθερο τόσες ημέρες για τους υπαλλήλους και όταν υπάρχουν ε, φερρυπίν ε, ημέρες άδεια επιπλέον για ταξίδι προς την χώρα προελεύσεως και από την χώρα προελεύσεως αναέτος τρεις και τρεις ημέρες, δηλαδή τρεις για να πάει ο υπάλληλος και τρεις για να γυρίσει. Συνολικά έξι ημέρες για να πάει στη χώρα του. Ποια είναι η τόσο δυσπρόσβατη χώρα της Ευρώπης για την οποία χρειάζεται τρεις μέρες ταξίδι κανείς. Να μου πει να πάω κι εγώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξηγήσω στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Πώς είναι δυνατόν να εξηγώ δηλαδή ότι υπάρχει σύστημα που επιτρέπει τέτοιε ακρότητε και ταυτόχρονα και τόσο υψηλού μισθούς. Δεν τα δικαιολογεί αυτά η η Επιτροπή. Δίνει κάποια απάντηση ως προς το πόσοι είναι οι υπάλληλοι της Επιτροπής που εισπράττουν πάνω από 10.000 ευρώ. και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν την, το χαμαλίκι όπως τα λέγαμε, τη βαριά δουλειά και κερδίζουν πολύ λίγα λεφτά. Βλέπουμε ότι είναι 7% οι πολύ χαμηλόμιστοι και πολύ υψηλό το ποσοστό εκείνων που κερδίζουν πάνω από 10.000 ευρώ. Η ερώτηση επίση, θα μείνουν τα πράγματα όπω έχουν, πώ προβλέπει την κατάσταση στην εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι υπενθυμίζω ότι εφέτο είχαμε νέο καταστατικό, άρα τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και μπρος η Επιτροπή και κάτι άλλο. Υπάρχουν 88 λειτουργικές θέσεις γενικών διευθυντών. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν 236 γενικοί διευθυντές στην πραγματικότητα. 236 άνθρωποι παίρνουν μισθό γενικού διευθυντή αλλά δεν κάνουν τη δουλειά του Γενικού Διευθυντή γιατί δεν είναι σε λειτουργική θέση Γενικού Διευθυντή όλοι τους. Από πού προκύπτουν όλοι αυτοί και γιατί. Και επίση για εμά ω αρχαίρμοδε για τον προπολογισμό, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε ε, να λειτουργεί ένα σύστημα το οποίο προβλέπει κάποιες θέσει που δεν είναι θέσει Γενικού Διευθυντή αλλά αμείβονται ω θέσει Γενικού Διευθυντή. Τρίτη ερώτηση. για την Κροατία. Υπάρχουν κάποιες θέσεις ε, εδώ μέσα στο μηχανισμό επαλήθευσης και προσπαθώ εδώ και χρόνια να καταλάβω τι έχουμε κερδίσει χάρη σε αυτό το μηχανισμό επαλήθευσης. Διότι βεβαίω φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συνεχίζεται η υποπτία, η παρακολούθηση ενό κράτου μέλου μετά και την είσοδο του διαφορετικά. Οι δυσκολίε ή αδυναμίε εντείνομαι πίστρο. Έχουμε λοιπόν εδώ την υπόθεση με τον κύριο Τούνσμαν, ο οποίο. είχε κάποιες ευθύνες σε σχέση με δημόσιους διαγωνισμούς και από εκεί πήρε κάποια χρήματα και ως εκ τούτου φαίνεται ότι είναι υπόλογος και φέρει ευθύνη. Υπάρχει λοιπόν κάποιος μηχανισμός ελέγχου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες. Δημόσιους διαγωνισμούς και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αναθέσεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε αρχές που διορίζονται και αφήνουν πεδίο ελεύθερο σε κάποιον κατά αυτόν τον τρόπο και ατιμωρητή να μπορεί κανείς να εισπράττει αυτά τα χρήματα. Τέταρτη ερώτηση και θα ήθελα γραπτή πληροφορία, ε, ενημέρωση παρακαλώ. Αυτό που μας είχε πει και ο κύριος Πίπαλξ. Για θέσεις του Ευρωπαϊκού Διαφορετικού Ταμείου για 977 συνολικά για το 2008, 997 συνολικά για το 2008, όπου δεν υπάρχει βέβαια ε, συμφωνία με τη βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε ορίσει ότι δεν πρόκειται να προσλάβει νέο κόσμο. Ποιος πήρε τις αποφάσεις αυτές στο... στην περίπτωση αυτή έχουμε πάλι και ζητήματα σφάλματο και θέμα σφάλματο από πλευρά του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ξέρω και από το Συμβούλιο ποιο ήταν αρμόδιο να κοιτάξει τα θέματα αυτά και να τα επαληθεύσει. Ευχαριστώ. Λέω πρώτος να ακούσουμε πρώτα κάποιες ερωτήσεις και μετά να απαντήσει η κυρία Ντέο. Ο κύριο Γκάιερ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. θα συμφωνήσω και θα συνεχίσω στα όσα είπε η κυρία Γκρέσλε με δύο ερωτήσεις. για τις οποίες δεν βλέπω να έχει λάβει απάντηση η Επιτροπή μας ε, από την Επιτροπή και την κυρία Τζέι. Για το χρόνο ταξιδιού δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε η κυρία Γκρέσλε νωρίτερα. Θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση νομιμότητα όλοι μα, όλα τα θεσμικά όργανα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει να κάνει και με την κακοπροαίρετη μερικέ φορέ παρουσίαση τη κατάσταση από τα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και από το γεγονό ότι μια φορά στα πέντε χρόνια καλούμε τον πολίτη να ψηφίσει στι ευρωεκλογέ, χωρί όμω να γνωρίζει τι κανόνε ισχύουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί ισχύουν αυτοί οι κανόνε. Όταν λοιπόν ένα υπάλληλο των ευρωπαϊκών ε, οργάνων που πληρώνεται το μισθό του χάρη στην εισφορά του Ευρωπαίου Φορολογουμένου. Έχει 7 μέρες διάθεσή του ανά έτος, προκειμένου να πάει στο χώρο καταγωγής του που ότι είναι δυσπρόσβατος και μάλιστα αυτό ισχύει για όλους, δεν είναι δυνατόν αυτό να το εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ζητήματα τα οποία εμείς ως Ευρωβουλευτές Και εδώ νομίζω δεν υπάρχει διάκριση ούτε μεταξύ υπαλλήλων επιτροπής, Υπαλλήλων Κοινοβουλίου ή Ευρωβουλευτών. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την υπόθεση της Ευρωπαϊκής αυτό δεν μπορεί δηλαδή να ισχύει για το Βέλγιο. Είναι δυνατόν να μου πείτε ότι θέλω τρει μέρε για να ταξιδέψω μέσα στο Βέλγιο ή στη Γερμανία, Φερρυπίν. Δεν υπάρχει, δεν νοείται τέτοια απόσταση. Μπε περιπτώσει υπάρχει μια τέτοια διάταξη, ένα τέτοιο κανόνα γενικό και πώ είναι δυνατόν να θεωρείται παραδεκτό κάτι τέτοιο. Εάν ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο, προφανώ ούτε στην επικοινωνιακή μα πολιτική ε, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό μπορούμε να ε, προβάλλουμε τέτοια επιχειρήματα. Όταν ε, τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, παραδείγματα, ε, εξετάζουν πόσα χρήματα κοστίζει ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα βγάζουν στη φόρα, θα ήταν καλό να έχω υπόψη και εγώ γραπτός πόσο κοστίζει η ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια. Γιατί ναι, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην έχετε πρόχειρα τα στοιχεία βέβαια στη διάθεσή σας, αλλά μπορώ να περιμένω μία γραπτή εξήγηση. Τρίτη παρατηρήση. Πώς μπορεί να καταλήξει η Επιτροπή σε μια δήλωση αξιοπιστίας αξιόπιστη και σχετικά σύντομα διότι έχουμε συζητήσει επί μακρόν την έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος. Εγώ όμως θα ήθελα να γνωρίζω πώς, σε ποιο βαθμό και σε ποιο πλαίσιο συζητεί το θέμα αυτό η, διαχείρι, η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τώρα δηλαδή είχαμε δει έναν ε, υπολογισμό ως προς την ε, οριακή χρησιμότητα των ελέγχων. Μπορώ δηλαδή να εξηγήσω εγώ σε έναν, ε, στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν ε, αξίζει να δαπανίσουμε 100.000 ευρώ φερρυπίν για να διορθώσουμε ένα σφάλμα που κοστίζει 0,5 ευρώ. Ναι, αυτό είναι λογικό και μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά πρέπει να έχουμε κάποια ιδέα του ποιο έλεγχο θεωρείται υπερβολικά δαπανηρός, υπερβολικά ακριβώ. και πώς διαπιστώνεται το ανεκτό περιθώριο σφάλματος ή ο ανεκτός, ο ανεκτός κίνδυνος σφάλματος. Ίσως θα ήταν ε, πιο σκόπιμο να έχουμε μια ανεκτή ποσόστοση ή ένα ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Ε, πριν γίνω ευρωβουλευτής δούλευα σε μια επιχείρηση και από εκεί έμαθα να εντοπίζω τον τομέα κινδύνου στον έλεγχο χρηματικών ροών ως εργαλείο διαχείρισης, ως βάση υπολογισμού. Και οφείλω να πω ότι ανησυχώ ως προς την ε, διατήρηση του όρου ανεκτός ε, κίνδυνο σφάλματος. Γιατί εν τέλει, εάν πρόκειται να, να είναι σε θέση να καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αξιόπιστη έκθεση αξιοπιστίας ε, και να προχωρεί πιο ε, απρόσκοπτα στην απαλλαγή, μπορεί αυτός ο ανεκτός κίνδυνος να φαίνεται ικανοποιητική λύση, αλλά δεν είναι επαρκής λύση. Και επανερχόμαστε στο πολύ ωραίο παραμύθι των αδελφών Γκριμ και τα ρούχα του βασιλιά, που όλοι έβλεπαν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά κάνει δεν τελμούσα να το πει. Αυτή είναι λοιπόν του ανεκτού κινδύνου σφάλματος, όπως έχει τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ακριβώς τα ρούχα, τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Όλοι λένε τι ωραία που είναι τα ρούχα, αλλά όλοι βλέπουν ότι ρούχα δεν υπάρχουν και ότι είναι γυμνός ο βασιλιάς. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει πια να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρίξω μια ματιά. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κ. Μόλτερ, η κυρία Ιβάνοβα, ο κ. Φιέλνερ και ο κ. Σοντή. Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Τέσσερις λοιπόν. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μόλτερ και μετά ας, δοθεί, ας δοθούν κάποιες απαντήσεις και μετά θα υποβάλουν τις ερωτήσεις οι υπόλοιποι τρία. Κύριο Μόλτερ, ευχαριστώ. Συντομότατο ερώτημα. Υπάρχει ένα σταθερό παράγον κάθε χρόνο στη συζήτηση, τα τελευταία 6-7 χρόνια επανέρχεται, οι αιτήσει εκθέσεις δραστηριοτήτων. Υπογράφονται από το Γενικό Διευθυντή για την ώρα και κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο ζητά στα ψηφίσματά του ο Επίτροπος να επίσης να υπογράφει. Και κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει όχι, δεν γίνεται αυτό, διότι ο Επίτροπος δεν μπορεί να υπογράψει. Θεωρώ ότι είναι απίστευτο που συμβαίνει αυτό. Γιατί μπορεί να υπογράψει επιστολή και να προβεί σε δήλωση στην Ελλομέλεια ο Επίτροπος να κάνει τα πάντα αλλά να μην αναλάβει ευθύνες για μια πολιτική που εφαρμόστηκε το προηγούμενο έτος και να υπογράψει μαζί με το Γενικό Διευθυντή. Πολιτική ευθύνη δεν αφορά το δημόσιο υπάλληλο, αλλά κάποιον που είναι υπόλογος προς το λαό. Και αυτός είναι ο επίτροπος. Εμείς πιθανότατα εκ νέου θα ζητήσουμε να συνυπογράφει ο Επίτροπος, ούτως ώστε εκείνος ή εκείνη να υπομισθούν τις ε, ευθύνες τους. Και πιθανότατα υποθέτω, και γι' αυτό θέλω απάντηση, Επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένας επίτροπος δεν μπορεί να συνυπογράφει τις αιτήσεις εκθέσεις ε, δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Γκράστα και ο κύριος Γκάιερ υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, λέγοντας ότι νομίζω ότι είναι θεμητό και ορθό ότι οι όροι απασχόληση όχι μόνο των ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι όλα τα θεσμικά όργανα έχουν κανονισμούς, τους ίδιους κανονισμούς για το προσωπικό. Είναι κανόνες που δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ενδείκνεται να λαμβάνεται υπόψη ότι η τεράστια πλειοψηφία του προσωπικού ζουν μακριά από τις πατρίδες τους και αυτό έχει κάποιες συνέπειες όσον αφορά το κόστος και τον 21ο αιώνα ακόμα υπάρχουν συνέπειες όσον αφορά το χρόνο για τα ταξίδια. Να σας δώσω εγώ κάποια δική μου εμπειρία, έτσι, ανακριτικά τα Χριστούγεννα. Οι πτήσεις μου ακυρώθηκαν και έπρεπε να οδηγήσω και να πάω στο Δουβλίνο. Μου πήρε 24 ώρες να πάω, 24 να γυρίσω. Ακόμα και με τι αεροπορικέ συγκοινωνίε τι σύγχρονε, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει κανεί στην πατρίδα του πάρα πολύ γρήγορα και γέρο για σημαντικέ ε, εκδηλώσει και γιορτέ, όπω τα Χριστούγεννα. Τούτου λεχθέντος νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα σε κάθε τομέα θέλει να βρει τρόπου βελτίωση, ότι οι κανόνε είναι σύγχρονοι, επίκαιροι. Στο προηγούμενο γύρο απαντήσεων ανέφερα ότι θα υποβάλουμε πρόταση για τη νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και εντό αυτού θα κάνουμε και στο διοικητικό κεφάλαιο κάποιε προτάσει για τον προπολογισμό και υποθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη ευκαιρία θα εξετάσει και το όλο θέμα των μισθών ε, και των επιδομάτων και τότε θα αποφασίσει κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να σας πω ότι δεν Αναγνωρίζω κάποια στοιχεία που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε και θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα ενδεχομένω για να τα καταλάβω καλύτερα. Δεν κατάλαβα το ότι 236 άνθρωποι πληρώνονται σε γενικοί διευθυντέ. Από πού το βρήκε αυτό, ταιριάζει με τα δικά μα νούμερα. σω αυτό θα έπρεπε διμερό να το ξεκαθαρίσουμε. Όσον αφορά το ευέλικτο ωράριο, ε, είναι πολύ σημαντικό η κοινωνική πολιτική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ένωση να ισχύει επίση και για το δικό τη προσωπικό και υπάρχει ένα σημαντικό θέμα συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής ζωή, και υπάρχει και το θέμα επίσης προσαρμογής των μεθόδων εργασίας που πρέπει να προσαρμόζονται στη σύγχρονη ζωή κυρίως το να μπορεί κανείς να ποικίλει να αλλάζει το χρόνο κατά τον οποίο εργάζεται. Χάρη στη βοήθεια τη σύγχρονη τεχνολογία, αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να δουλέψει κανεί σε διαφορετικέ χρονικέ περιόδου και να αποδίδει κατάλληλα και νομίζω από την, ε, την όλη κουλτούρα της παρουσίας θα κινηθούμε στην κουλτούρα ε, των αποτελεσμάτων. Θέλουμε τον ευέλικτο ωράριο να εφαρμόζεται σύγχρονη όρια εργασία στο προσωπικό μας. Έδωσα αριθμούς και στοιχεία και νομίζω προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια σύγχρονη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού, το management. Όλοι θα γνωρίσετε τι επαφέ σα με προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι που ξεπερνούν κατά πολύ το ελάχιστο ωράριο εργασία την εβδομάδα και αυτό διότι είναι αφοσιωμένοι στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Και κάποιο θα πρέπει να έχει ε, την αίσθηση τη αναλογία όταν εξετάζει αυτά τα θέματα. Τώρα τα όσα είπε και ο Σπίμπαγκς, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό κυρία Γκρέσλε, δεν έχω τις πληροφορίες πρόχειρες, με τα χαράς να σας απαντήσω γραπτός. Όσον αφορά τον ανεκτό, τον ανεκτό ποσοστό κινδύνου, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το συζητήσαμε με το ελεκτικό συνέδριο που το επεξεργάστηκε πολύ το θέμα και έκανε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστεί αυτή η έννοια δεν πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να καθορίσουμε τον ίδιο αριθμό, το ίδιο ποσοστό σε κάθε τομέα πολιτική, γιατί διαφέρει κάθε τομέα, όπω η κοινή αγροτική πολιτική, είναι μια κοινή πολιτική, δικείται κεντρικά, η πολιτική συνοχή είναι αποκεντρωμένη με κοινή διαχείριση. Και αυτό που συζητούμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι θεωρούμε εμείς ότι είναι το ενδεδειγμένο ποσοστό κατά τομέα πολιτικής και θα υποβάλουμε λεπτομέρειες είναι θέμα της σωστής ισορροπίας, της σωστής αναλογίας. Δηλαδή θέλουμε από τη μια να έχουμε αποδεκτό ποσοστό κινδύνου και από την άλλη αποδεκτό επίπεδο ελέγχου. Αλλά κατά την άποψή μου δεν θα είναι τα ίδια ποσοστά σε κάθε τομέα πολιτικής. Έχουμε καταποκοπή ποσό 2% για την ώρα, το ποσοστό αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι είναι το σωστό ποσοστό γενικά και υπάρχει περιθώριο για συζητήσεις και όταν θα ολοκληρωθούν οι συζητήσει εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα χαρά να μοιραστούμε την ανάλυση και τη λογική που θα ακολουθήσουμε για να προτείνουμε διαφορετικά ποσοστά σε διαφορετικού τομεί πολιτική. Αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα να συζητηθεί με την Επιτροπή σα, με το Λεκτικό Συνέδριο, με τα χαρά να συζητήσουμε. Ε, ήδη όσον αφορά το ερώτημα του κ. Μόλτερ για τι ετήσει τι εκθέσει δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό ο Γενικό Διευθυντή να υπομειστεί τι ευθύνε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τη μοιραστεί με κάποιον άλλον. Είχαμε ένα θολό σύστημα πριν που μα οδήγησε σε δυσκολίε. Είτε μπορεί να έχει κανεί πολιτική ευθύνη με τον κεντρικό έλεγχο και τη βαριά γραφειοκρατία που αυτό συνεπάγεται, είτε αποκεντρωμένο έλεγχο όπου οι γενικοί διευθυντέ είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι που διαθέτουν, στη διάθεσή του. Αυτό δεν απομακρύνει την πολιτική ευθύνη, τη συλλογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συλλογικά επομίζεται ε, την πολιτική ευθύνη για τις ε, αιτήσει εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να αναμίξει κανείς στοιχεία διαφορετικών συστημάτων και ούτω τρόπος ε, τάχιστα θα αντιμετωπίζαμε δυσκολίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα πάμε σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων τώρα τρεις συνάδελφοι του ΕΛΚ, η κυρία Ιβανόβα, ο κύριος Φιέλνερ και ο κύριος Οντί. Εγώ θα προσέχω την ώρα, το χρόνο. Δύο-τρία λεπτά ο καθένας. Η κυρία Ιβάνοβα πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής ήδη αναφέρθηκε στα σημαντικότερα ζητήματα και ερωτήματα που ήθελα να θέσω όσον αφορά τα συστήματα ελέγχων και την ποιότητα των στοιχείων και η κυρία Ντέι ανέφερε ότι έγιναν πολλές βελτιώσεις ευπρόσδεκτες. Όμως έχω κάποιες ερωτήσεις. Παραδεχόσαστε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αδυναμίες οι οποίες θα έπρεπε να ξεπεραστούν τόσο ώστε να βελτιωθεί ο έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των κρατών μελών σε την ποιότητα των στοιχείων των ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων και πού ακριβώς διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αδυναμίες. Πέρα από τη συνοχή που αναφέρατε και την πρόθεση να εισαχθούν κάποια συμβάσεις με τα κράτη-μέλη για να αυξηθούν οι ευθύνες που επομίζονται ε, και άλλες ερωτήσεις που αφορούν την Κροατία και την Μακεδονία, λέει ο Μιλήτρια. Για την Κροατία αφορά τα επίπεδα τους φακέλους που απορρίπτονται και επιστρέφονται στις χώρες. Είναι ικανοποιημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το 20% ποσοστό απορρίψεων για την Κροατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Κροατικές Αρχές τι κάνουν για να μειώσουν περαιτέρω το ποσοστό. Και για το θέμα Τούσμαν στην ε, Κροατία, λέει και η κυρία Γκρέσλε, για τη Μακεδονία, λέει ομιλήτρια, καθιστές τη διαδικασία χορήγηση στο ΦΥΡΟΜ ενός εργαλείου διαχείριση και αναμένεται αργότερα, πιθανότατα το 2010, λέει ο Μιλήτρια, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η πρόοδος ε, σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε υπενθυμίζει ένα ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Ιβάνοβα όσον αφορά τον κ. Τούτσμαν Ίσως αυτό θα μπορούσατε να το απαντήσατε. Ο κ. Φιάλνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντέ για τις γραπτές της απαντήσεις. Παρέχονται πολλές καλές πληροφορίες. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απαντήσεις που δόθηκαν. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα ε, το χρόνο εργασίας και πόσος χρόνος χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς από το α στο β Α, τα αφήνουμε αυτό για την κυρία Γκρέστα για μελλοντικέ συζητήσει, διότι αυτό θα μου έπαιρνε το χρόνο μου. Για τα δύο λεπτά. Για τι εθνικέ δηλώσει τώρα. Έχουμε κάποια πρόοδο εκεί και νομίζω ότι είναι καλό να το επαναλαμβάνουμε και να το λέμε αυτό, διότι συχνά εκεί στην Επιτροπή αυτή θεωρεί κανεί ότι κάθε χρόνο, κάθε χρόνο τίθεται τα ίδια ερωτήματα και φαίνεται ότι δεν προχωρούν τα πράγματα. Είναι πολύ καλό να βλέπουμε ότι καμιά φορά πετυχαίνουμε κάποια πράγματα και αυτό είναι καλό. Αυτό όμως που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθά ποικιλοτρόπως τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις. Κατά κάποιο τρόπο είναι καλό ότι απάντηση στην επιστολή από Ολλανδία και Σουηδία θα καταφτάσει ίσως κάπως καθυστερημένα αλλά διαβάζοντας την απάντησή σας τι με εξέπληξε ότι ε, ζήτησαν καθορισμό βασικών πτυχών για τι εθνικέ δηλώσει. Και αυτό που απαντήσατε, που θα δώσετε, ίσω δεν το κατάλαβα καλά. Λέτε, θα τους δώσετε όμως, προσανατολισμό για τα χαρακτηριστικά όσον αφορά την η αξία. Το σημαντικό ποιο είναι, να γίνουν συγκρίσιμα τα στοιχεία. Και θα ήταν θλιβερό αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα εκεί, αν υπάρξει εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη δεν την χάνουν της υποστήριξης που θα ήθελαν όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις. Κάτι θέλαμε και εμείς. Πρώτο ερώτημα ήταν αυτό. Δεύτερο, πειθαρχικές δράσεις. Στη γραπτή σας απάντηση λέτε ότι είχατε νέα υποθέσεις που οδήγησαν σε έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι καλά μαντάτα. Πολλοί εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο εννέα ίσως να είναι καλό, κακό, τι να πω, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Αλλά καταρχάς θα ήθελα να καταλάβω, πειθαρχικές διαδικασίες, τι σημαίνει αυτό. Είναι το ίδιο με δράση, θα σημάνει δράση κάτι τέτοιο. Ή θα έχουμε εννέα διαδικασίες και δύο καταλήξουν σε κάποιες πειθαρχικές δράσεις. Και θα καταλάβω ποια είναι η κοινή δράση, τι είναι η κοινή δράση, ποια είναι η κανονική πειθαρχική δράση, η συνήθις πειθαρχική δράση σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν μπορούσατε να μου δώσετε κάποια απάντηση πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σοντή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Θέλω να του πω πραγματικά ότι είμαστε πολύ τυχεροί να ακούσουμε ε, τις παρατηρήσεις του και την ενέργεια που τον έχουμε να μας δίνει τόση ενέργεια. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις έχω να πω κάτι. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο. Δηλαδή, όταν ζητάμε από τα κράτη και από τους υπουργούς να μας λένε πιστοποιήστε, ο, πιστοποιήστε μου ότι είναι καλή η λογαριασμοί, αυτό δεν είναι δική του δουλειά, είναι του ελεκτικού συνεδρίου. Αν εν ονόματι ελέγχου του ζητούμε να μα επιβεβαιώσουν ότι έχουν διαθέσει τα πάντα, ότι οι εθνικές αρχές ελέγχου είναι ανεξάρτητε, ειδού ε, ο υπουργό θα πρέπει να τοποθετηθεί. Προτείνω να παραμείνει αυτή η έννοια, να επεξεργαστούμε όμω το περιεχόμενο τη δηλώσεως αυτή της δηλώσης αξιοπιστίας. Όσον αφορά τη διαδικασία τη γενική, εδώ και 16 χρόνια συζητούμε το θέμα. Εγώ θέτω το ερώτημα στο ελεκτικό συνέδριο. Ναι ή ου έχουμε μια δήλωση αξιοπιστίας. Ο εισηγητής λέει έχουμε δήλωση αρνητική αξιοπιστίας. Εγώ δεν τη βλέπω. Η συνθήκη ζητά από το ελεκτικό συνέδριο να δώσει μία δήλωση αξιοπιστίας. Όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, και σε όλε τι ε, υποκείμενε συναλλαγέ. Όσον αφορά εξοπιστία των λογαριασμών, έχουμε επιστοποίηση ανεπιφύλακτη. Όσον αφορά τι υποκείμενε συναλλαγέ, το Ελεκτικό Συνέδριο ε, δίνει γνωμοδοτήσει. Δύο θετικέ και οκτώ αρνητικέ τοποθετήσει. Δεν είναι όμω δήλωση. Μία δήλωση. Θα ήθελα να ξέρω αν ναι ή ου έχουμε δήλωση αρνητική ή ενδεχομένω είναι θετική. Και ποια είναι η δήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την εφαρμογή ε, των συνθηκών. Όσον αφορά τα όσα είπε η κυρία Γενική Γραμματεύς, μπορείτε να μας πείτε τίποτα για τις σχέσεις με το Συμβούλιο, διότι στην Κοκομπίου Συχνάκης διεξάγονται συζητήσεις όσον αφορά άρνηση απαλλαγής παραγματος χάρη, που δεν είχε πάρα πολλές συνέπειες πολιτικές, όσον αφορά το Συμβούλιο, άρνηση απαλλαγής. Με τους συναδέλφους σας, γενικούς γραμματείς του Συμβουλίου, έχετε σχέσεις, διότι πάντα εκπλησόμην από τις κακές σχέσεις που υπήρχαν με το Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Εσείς που ουσιαστικά είσαστε υπεύθυνοι για την ε, γενική ενοποίηση των ε, λογαριασμών. Ενώ το ελεκτικό συνέδριο δεν κάνει καμία παρατήρηση ελάχιστον αφορά τη διαχείριση του Συμβούλιου. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Έχω εγώ μια ερώτηση. Θα ήθελα να θέσω. Η απάντηση που δώσατε, κυρία Γενική Γραμματεύς, στο ερώτημα 1 όπου είπατε ότι τίθεται το θέμα των εθνικών λογαριασμών. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβησε κάποια ανάλυση και σύντομα θα στείλουμε κάποια κατευθυντήρια, κατευθυντήριο σημείωμα. Το ερώτημά μου είναι, αυτή η ανάλυση είναι διαθέσιμη, είναι στη διάθεσή μας, μπορεί να διαβιβαστεί στον εισηγητή, στο βασικό εισηγητή. νομίζω ότι θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον λοιπόν αυτό ε, να μας δώσει κάποιες ε, ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και είπατε ότι σύντομα θα αποσταλεί ένα σημείωμα κατευθυντήριο με κατευθύνσεις. Ε, τι εννοείτε με σύντομα, πότε θα συμβεί αυτό. Λοιπόν... Ε, Πώς το ακριβώς το χρόνο. Έχετε το λόγο τώρα παρακαλώ κύριε Τζέι. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω με τη σειρά στις ερωτήσεις, καταρχάς στι εθνικές δηλώσεις θα πιέζουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν και τι συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να, να συμφωνήσουμε τι εννοούμε και ποιος έχει την ευθύνη για την ε, υποβολή των αιτήσεων. Κατά τα άλλα μπορούμε να σε υποστήλουμε μια σύντομη ανάλυση στην οποία έχουμε ήδη προβεί των αποτελεσμάτων και τη αποδοτικότητα ορισμένων μέτρων στα οποία έχουν προβεί τα κράτη-μέλη που έχουν προχωρήσει στον δρόμο αυτό. Και όταν λέμε κατευθυντήρε γραμμέ, εννοούμε όντω ότι θα καθοδηγούμε τα κράτη-μέλη όταν αυτά θέλουν περισσότερο η εναρμόνιση και η χρονική και ω προ το περιεχόμενο. Γιατί και η χρονική στιγμή κατά την οποία κατατίθενται αυτέ οι δηλώσει έχει μεγάλη σημασία για να κλείνουν οι λογαριασμοί καθ' έτου κτλ. Ω προ τι πειθαρχικέ διαδικασίε. Καταρχά, πριν να γνωρίζουμε εάν ε, κάποιος θεωρείται πως έχει παραβιάσει τους κανόνες, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία. Πάντοτε ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Δεν μπορώ λοιπόν να σας ε, προ... Ε, αναγγείλω πόσες από αυτές τις πειθαρχικές διαδικασίες θα καταλήξουν σε κυρώσεις. Υπάρχουν όμως κυρώσεις, δυνάμει του κανονισμού προσωπικού, εφόσον κάποιος αποδειχθεί ότι έχει παραβιάσει τον κανονισμό, κυρώσεις είτε η απώλεια βαθμού ε, μέχρι την ε, απόλυση για τις πολύ σοβαρές περιπτώσεις και παραβιάσεις. Μας περιπτώσει, οι από τις περιπτώσεις ε, έχουν να κάνουν με μία επαγγελματική συμπεριφορά, με παρενόχληση, μερικές φορές με οικονομικά ζητήματα, φερρυπίν, δηλώσεις δαπανών κτλ. Ε, λίγο πολύ έχουμε το ίδιο φάσμα προβλημάτων που θα εντοπίζονταν σε οποιοδήποτε αντίστοιχη μεγάλη ομάδα ατόμων. Ας προς σχέση σχέσεις με το Συμβούλιο. Ναι, συζητώ τακτικά και με τους ομολόγους μου του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αρκετές φορές το χρόνο όλοι οι γενικοί διευθυντές όλων των θεσμικών οργάνων συναντώνται για να συζητήσουν θέματα πολιτικής και κοινά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, τη διοίκηση κτλ. Πιέζουμε το Συμβούλιο και τα κρατημέλη βέβαια και τη Γραμματεία για όλα αυτά τα θέματα και τις εξελίξεις. Νομίζω ότι μας ε, κοιτούν με καχυποψία γιατί θεωρούν ότι είμαστε πολύ κοντά στο Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν σπέβδουν με περισσή χαρά να υλοποιήσουν τα όσα τους ζητούμε, αλλά βάσει όπως εμείς εξακολουθούμε να τους πιέζουμε και πιστεύω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσφατη δημιουργία τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Φερρυπίν ήταν μια στην οποία συνεργάστηκα στενά με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, διότι ήμασταν και οι δύο στρατευμένοι στην υπηρεσία αυτή, στην, στον αγώνα δηλαδή να δώσουμε νέο προσωπικό από το δικό μα προσωπικό στην υπηρεσία αυτή, αλλά ταυτόχρονα και να προσδιορίσουμε όλου του κανόνε ε, για τη στελέχωση κτλ. Άρα μπορεί να συναντηθούμε και εκτός των προγραμματισμένων ε, ε, συνεδριάσεων όταν υπάρχει ανάγκη. Και βεβαίως και με το Γενικό Γραμματέα του ε, Κοινοβουλίου πολύ πιο τακτικά από ό,τι με τους άλλους φορείς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο δεν έχει ε, απαντηθεί, δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση Τούτσμαν, για τον Τούτσμαν. Κυρία Γκρέσλε, κάντε μου τη χάρη. Έκανα λάθος. Ο Σανάντερ ήταν πρόεδρε, όχι ο Τούντσμαν. Λάθος έκανα. Η Ιλιάνα ε, επίσης από ό,τι φαίνεται δεν έλαβε απάντηση στην ερώτησή της για την Κροατία. Φαίνεται ότι η Κροατία είναι αγαπητό θέμα πάντοτε. Έχετε την καλοσύνη κυρία Ντέι. Απάντηση. Ε, δεν μπορώ να σα δώσω συγκεκριμένη ερώτηση ούτε για την Κροατία ούτε για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Θα ήθελα απλώ να επισημάνω ότι θα έρθω σε επαφή με του αρμόδιου γενικής διευθύνσεως για τη διεύρυνση και να σα καθασυχάσω ότι για την ε, ταξιακή διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τι αρχέ τη ψήφιας για ένταξη χώρα, χώρας ώστε σταδιακά να εξασφαλίζεται πω ε, θεσπίζονται όλοι οι θεσμοί, οι δομές, οι, ελεκτικές, ε, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, ώστε όταν έρθει η ώρα για ανάληψη από την λόγω χώρα του, της διαχείρισης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πλήρως έτοιμη όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Πρόκειται βεβαίως για προσαρμογή φυσταμένων μηχανισμών ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους δικούς μας κανόνες κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι όταν βλέπω κάποια ποσοστά αποτυχίας, αλλά πρέπει να πω ότι όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά ή μάλλον απόρριψη αιτήσεων, φαίνεται ότι αυτό ε, επαληθεύει πως το σύστημα λειτουργεί καλά. Έστω και αν δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, τηρούνται οι κανόνες. Πάντως, για πιο πολλά ε, στοιχεία, πολύ ευχαριστώ να σας στείλω γραπτός απαντήσεις για τις δύο χώρες. Κυρία Γκρέσλε, μα, θα ήθελα να μου πει, ε, εδώ στον κύριο, με το περίπτωση του κυρίου Σανάντερ, πρόκειται για κρατική εγκληματικότητα, για εγκληματικότητα καθαρή. Ο πρόεδρος, θα μείνουμε σε αυτά δεδομένες κατάστασης. Ο κύριος Οσί, κύριο, ο κύριος Οντή, αναφέρθηκε σε εσά κύριο Οσί, υπάρχουν ερωτήσεις για το ελεγκτικό συνέδριο, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για τον κύριο Οντή, λοιπόν, και τα σχόλιά του. Θα ήθελα να παραπέμψω στην κυρία Κάλλη για την απάντηση. Αυτή είναι η αρμόδια για την ε, έκθεση αξιοπιστία. Όταν έρθει η ώρα να τη δείτε στην Επιτροπή, σα παρακαλώ να επιτρέψετε να σα απαντήσει εκείνη. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω τα εξή. Έχουμε να κάνουμε καταρχά με την αξιοπιστία των, ε, της στηρίσεως των λογαριασμών. Άρα γίνεται μια αξιολόγηση όπου λέμε ότι όντως οι λογαριασμοί αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές τις οποίες παρουσιάζουν. Δηλαδή είναι πραγματικέ συναλλαγέ. Και επίση, στη γνώμη μα, στη νομοδότησή μα, δίνουμε και στοιχεία σχετικά με την νομιμότητα, το σύνομο των πράξεων αυτών. Και σημειώνουμε εάν θεωρούμε ότι υπάρχουν σφάλματα όπως προς κάποιες δαπάνες σε ουσιαστικό. Εκεί λοιπόν περίπου έχουμε 2% σφάλματος εντοπίσει. Και εδώ πρόεδρε σας, παραθέτω, σας παραπέμπω στις σελίδες 11 και 12 του πρώτου κεφαλαίου της ετήσιας εκθεσής μας. Αλλά αν επιτρέπετε κυρία Κάλλη τον έρθει να σας δώσω τα πιο τεχνικά στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Χατζημαρκάκης παρακαλώ να κάνει ακόμη μερικές παρατηρήσεις για να προχωρήσουμε, να πιάσουμε το θέμα αυτό στην Ο κύριος Χατζημαρκάκης, κύριε Αντέ, με χαρά σας ακούω. Δώσατε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Και δώσατε απάντηση κατανοητή. Τα καταλαβαίνω όλα όσα είπατε δηλαδή. <laughs> Όχι, και αυτό κέρδος είναι, μη λέτε. Ωστόσο, σε ένα βαθμό μου έχετε ζωγραφίσει τα πράγματα πολύ ρόδινα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, επιτεύγματα υπάρχουν, ναι, προσπάθειες υπάρχουν, γίνονται. Ξέρω ότι κι εσείς είστε ευγνώμων από την πλευρά σας για τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σας βοηθούν έτσι. Αλλά αρκούν όλα αυτά. Ως προς το ερώτημα που υπέβαλα νωρίτερα για, την εξωτερική, ε, για τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο. Είπατε ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος και ότι είναι αυτό αρμόδια αρχή για το εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο. Ναι, ωραία. Τη λαμβάνω αυτή την υπόθεση λοιπόν, την καταγράφω, σας λέω ναι ευχαριστώ για την απάντηση, σωστή απάντηση, αλλά σας δίνουν αρνητική έκθεση αξιοπιστίας από το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι σαφέστατο αυτό στις δύο-τρεις σελίδες ότι η δήλωση είναι αρνητική. Εσείς όμως μου λέτε ότι τη δέχεστε την αρνητική δήλωση αξιοπιστίας χωρίς δυσκολία, διότι καταβάλλετε τις προσπάθειές σας και βελτιωνόσαστε. Αυτό μας είπατε και αυτό κατανοητό. Αλλά δεν αρκεί, θεωρώ. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω τους στόχους της πρώτης Επιτροπής Βαρόσο, που στόχο είχε την θετική έκθεση αξιοπιστίας. Και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ευκαιρία δοθήσει να ασκήσουμε περισσότερε πιέσει σε εκείνου που σα προξενούν τι δυσκολίε. Και αυτοί είναι τα κράτη-μέλη. Δεν είστε εσεί οι ίδιοι, αλλά τα κράτη-μέλη. Εν πάση περιπτώσει, τα σχέδια δράση καλά είναι, δεν αρκούν όμω. Μα λέτε επίση ότι θα πρέπει να συνεργάζεστε με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλιστούν κάποια επίπεδα, κοινά επίπεδα. Ναι, γίνεται ε, προοδό και από άλλου επιτρόπου. Φερρυπίν σε μια ακρόαση με την κυρία Ανδρούρα Βασιλείου, που ήταν η πρώτη φορά όπου προσεκλήθη η Επίτροπο Αρμόδια για την εκπαίδευση στην Επιτροπή μα και εξεπλάγει. Τη άρεσε όμω η ιδέα, διότι δεν έχει τίποτε να κρύψει. Και δισετησίω οργανώνει ε, σεμινάρια με τα αρμόδια σε εθνικό επίπεδο όργανα για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Δισετησίω λοιπόν σεμινάρια, τεχνογνωσία, ε, εξηγούν τι πρέπει να γίνεται κτλ. Βέλτιστη πρακτική αποτελεί αυτό. Και αναφέρομαι σε μια άλλη γενική διεύθυνση, ε, χαρτοφυλάκιο άλλου επιτρόπου που κάνει εξαίρετη ε, δουλειά. Όμως η Γενική Διεύθυνση για, την περιφέρεια, για τις περιφέρειες και το κοινωνικό ταμείο βλέπουμε ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Οι πρακτικές τους δεν είναι ικανοποιητικές Και πρέπει να σταματήσει αυτό. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρός σας, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαρόσο, ερωτώμενος σε επίπεδο ε, στην όλη μέρα του Κοινοβουλίου στις 14 Δεκεμβρίου του 2010 για τα κράτη-μέλη έδωσε την εξής απάντηση. Η ερώτηση ήταν τι μπορεί να πράξει για να βελτιώσει τις επιδόσεις των κρατών μελών. Εντός παρενθέσεως βέβαια, η ευθύνη δική σας είναι οι επιδόσεις των κρατών μελών. Κλείνω η Απαντά λοιπόν ο κύριος Μπαρόσο. Όσον αφορά την, την ερώτηση σας, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ε, πλην των 4-5 εκείνων κρατών μελών. Αυτό μιλά αυτό αναφέρεται στην εθνική δήλωση, τα οποία δεν είναι έτοιμα για την υποβολή τη εθνική δηλώση αξιοπιστία. Και αληθεύει όντω αυτό που είπε ο Γενικό Διευθυντή, ότι δεν είναι στη διάθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε όλα τα απαραίτητα μέσα για να ε, εμπλακεί ε, στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη το νωρίτερο δυνατό και να επαληθεύει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται σε εθνικό επίπεδο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Άρα, ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκάθαρα λέει ναι, δεν έχουμε, στη, δεν έχουμε στη θέση μας τα στοιχεία μας που χρειαζόμαστε, αλλά τα λεφτά τα δίνουμε. Και εσείς μου λέτε ότι αυτό σας φαίνεται εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Αυτό σας λέμε και εμείς. Και δεν είναι εντάξει να σας λέει το ελεγκτικό συνέδριο 30% κακώς κατεβλήθησαν και να το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλευρά Και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε εις βάθος όλο αυτό το πράγμα. Πότε θα έρθει η μέρα που θα σταματήσει αυτή η πρακτική. θα συνεχίσουμε την πρακτική την οποία ανακάλυψαν και συζήτησαν και κάποιοι συνάδελφοι εδώ βήμα προς βήμα. Ναι, είναι μία λύση ενδεχομένως προσωρινά, αλλά τώρα πρέπει πια να κάνουμε το άλμα που σημαίνει να γυρίσει ο τροχός και να γυρίσει ο τροχός στην ορθή κατεύθυνση. Κάποια κρατημέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προφανή οικονομική κρίση, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία ε, λαμβάνουν πολλά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και αν συνεχίσουμε τα χρήματα αυτά να τα διαθέτουμε κατά τον τρόπο που, τα διαθέτουμε, δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουμε τι χώρε αυτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να κλείσουμε το χάσμα συνοχή μεταξύ των πλουσίων και των μη πλουσίων κρατών. Γιατί αυτό είναι ο στόχο μα. Ο στόχο μα δεν είναι να ε, του ε, καλλιεργήσουμε αυτή την ε, νοοτροπία του δικαιούμε ε, χρηματοδότησης. Ε, αυτή η νοοτροπία πρέπει να σταματήσει. Και αυτό θα το εξασφαλίσουμε με σαφείς στόχους που θα εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη, θα τους δείξουμε ποια είναι η προστέμενη ασυξία σαν πρώτο βήμα και επίσης θα πρέπει να αναλυθεί το τι έχουν πράξει τα κράτη-μέλη, πού έχουν υπογράψει και ποιο στις συμβάσεις. Και σας διαβεβαιώ ότι βεβαίως θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας. Σας διαβεβαιώ ότι θέλουμε ένα πρόγραμμα δράσης από πλευρά σας για τη μέθοδο χάρη στην οποία θα καταστούν πιο υπεύθυνα τα κράτη-μέλη όταν υπογράφουν τη σύμβαση. Αυτή η ιδέα των συμβάσεων είναι πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα. Αν μπορούσατε περισσότερο να την αναπτύξετε, έτσι ώστε να μας παρουσιάσετε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς σκοπεύετε να την υλοποιήσετε, θα ήταν πολύ καλά. Βεβαίως όμως παρακαλώ να μην λησμονήσετε και την άλλη υπόθεση. Την ανάκτηση των αχρεωσίτων καταβληθέντων. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε στον φορολογούμενο 7,8 δις χαθήκαν διαπαντός. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και ελπίζω ότι θα έχουμε και στο μέλλον αγαστή συνεργασία και τι, και τι ορισμένες φορές δύσκολη. Πάντως πιστεύω ότι το σπρώξιμο το δικό μας είναι καλύτερο από το να μην υπάρχουν οι πιέσεις που υφίσαστε από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ντέι για την παρουσία της, για το πνεύμα συνεργασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, μας απασχολεί όπως βλέπετε. Κυρία μου, το βλέπουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Εδώ και μια μισή ώρα το συζητούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της εκθέσεως που θα υποβάλει ο κ. Χατζημαρκάκης και είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί και συνέχεια στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ και περνούμε στην απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Η συγκητή είμαι εγώ και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διακοπή για να δώσουμε το την προεδρία στον κύριο Οντζή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση με το σημείο 8 της μερικής διάταξης. Μάλλον θα πρέπει να αφήσω λίγο περιθώριο χρονικό για να τελειώσουν οι συνομιλίες. Σημείο 8 στην εμμυρή Διάταξη. Απαλλαγή 2009. 8ο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, λέει ο Πρόεδρο. Χαιρετίζω εδώ την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκπροσωπούμενη από τον κύριο Τάμσιν Μπάρτον, Γενικού Διευθυντή για τι Δραστηριότητε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν. τη κυρία, κυρία Μπάρτον είστε. Είστε κυρία, με συγχωρείτε. Στα χαρτιά μα είναι κύριος. Βλέπετε ότι κακώ δεν σα συναντιάμε πιο συχνά και δεν σα γνωρίζουμε. Υποβάλλω λοιπόν τη συγγνώμη μου κυρία μου και παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να με λέτε δόκτωρα Μπάρτον, άμα ε, θέλετε. Έτσι δεν θα υπάρχει και πρόβλημα να καθορίσετε το φίλο μου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε. Όταν ήμουν γενική Διευθύντρια για τις εξωτερικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, ήρθα στην τράπεζα τα μέσα, στα μέσα Νοεμβρίου. Ε, είμαι λοιπόν στην αρχή και χαίρομαι γιατί θα μπορέσω να ακούσω κάποιες καλές ιδέες από τις ερωτήσεις που θα μου θέσετε σήμερα. Αυτά από πλευρά. Ο λόγος εισηγητή, λοιπόν, ο κύριος Μπάρτης Θάης. Ehm, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που είναι εδώ εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και που είναι εδώ και η κυρία Μπάρτον. διότι είναι αρμόδια εντός της τράπεζας ε, με, για τις δραστηριότητες με τρίτες χώρες, με χώρες ΑΚΕ. Κατά την προετοιμασία της συζήτησης και κατά την προετοιμασία της συζήτησης που κάναμε πριν από δύο εβδομάδες με τον Επίτροπο Πίμπαλξ, χρησιμοποίησα τα ψηφίσματα για την απαλλαγή των τελευταίων τριών-τεσσάρων ετών. Όπως έλεγα πριν από δύο εβδομάδες και στον Επίτροπο Πίμπαλξ, διαπίστωσα ότι κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια όταν συζητά την απολογή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και κυρίως τα θέματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Όσον αφορά, δεν θα έλεγα τόσο τις δυσκολίες, αλλά τις δυνατότητες που έχουμε εμείς ως αρχή ελέγχου του προϋπολογισμού, έχουμε πάντα λοιπόν κάποιες δυσκολίες και δεν έχουμε μια τόσο σαφή εικόνα. Η δήλωση, δήλωση αξιοπιστίας δεν αφορά τα κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε αγαστές σχέσει και μια καλή ετήσια έκθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κυρίως όσον αφορά τα μέσα επενδύσεων. 3,4 δι διακυβεύονται εδώ και ε, προκύπτουν από την απαλλαγή, αλλά είναι δημόσια κονδύλια τα οποία καταβάλει ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος. το πλαίσιο που έχουμε δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα χρήματα και κυρίως τι αποτελέσματα επιτυγχάνουμε. Ε, σαφώς η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μας δίνει αρκετές πληροφορίες, αλλά αυτές οι πληροφορίες είναι χρηματοοικονομικές και δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορίες ως προς τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται. Να καταλάβουμε δηλαδή πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς επιτυγχάνεται. σε όλα τα ψηφίσματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και η Ολομέλεια ζητά περισσότερες πληροφορίες ως προς τα αποτελέσματα. διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή και τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στα πέντε ερωτήματα που θέσαμε. Κάποια εξ αυτών ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα και ε, βασίστηκαν και στα όσα ανέφερε ο τύπος ε, και μάλιστα νομίζω ότι συνέπιπτε και χρονική περίοδος με τη δική σας ανάληψη καθηκόντων. Ε, είχαμε κάποια άρθρα στην Guardian τότε τα οποία προέκυψαν από την ε, έρευνα που έκανε η μη κυβερνητική οργάνωση Count Balance. Και διαβάζοντας τις απαντήσεις σας, ε, καταλαβαίνουμε και σε τι πλαίσιο εμπίπτουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις απαντήσεις σας. αλλά σε κάποιο σημείο στις απαντήσεις που μας δίνετε, ε, κυρίως ε, για την ερώτηση 5, την οποία θα ήθελα να αναφέρω εδώ, Μας λέτε και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συγγνώμη για αυτό το πέρα δόθε, ψάχνω να βρω και πού ακριβώς είναι το κείμενο. Διαβάζω στα αγγλικά. Όλες οι πληροφορίες που διατίθεται από την πληροφορία μπορούν να δοθούν κατόπιν ετήσεως, εκτός και αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικέ. Η φράση στα αγγλικά είναι compelling reasons for non-disclosure. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λόγοι που μπορεί να μην μας επιτρέπουν να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες ή να διαθέσουμε αυτές τις πληροφορίες η διαφάνεια είναι υψής της σημασία σε αυτή την περίπτωση. Στην απάντηση λοιπόν που δίνεται στην ερώτηση υπ. 5, σε κάποιο σημείο αναφέρεστε και σε διάφορες μορφές απάτης που διαπιστώθηκαν. Στη σελίδα 11 εκ των 17, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λέει βάσει συγκεκριμένων δικλείδων δασφαρίας ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης ε, προς το συμφέρον της ε, κοινότητας και της περιοχής έχουν δημοσιοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή και στην Όλαφ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Ποιες είναι αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις απάτης που αναφέρονται εδώ. Και επίσης Πού τις διαπιστώσετε, τι ποσά αφορούν, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες του Γενικού Επιθεωρητή και της Όλαφ. Έχουμε επιτύχει κάποια αποτελέσματα. Τέλος πάντων, πώς έχει η κατάσταση. Στην απάντησή σας, για μια ερώτηση που είχαμε για τη μαύρη λίστα και το ποιους περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα, λέτε ναι έχουμε καθορίσει κάποιες πρακτικές, κάποιες πρακτικές οι οποίες συνάδουν ε, με τα όσα ε, γίνονται και τους προσανατολισμούς που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι για τη μαύρη λίστα. Ποιους μαυροπινακίζουμε και για ποιο λόγο, κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Επίσης, ε, σε όλα τα ψηφίσματα που έχουμε για την απαλλαγή που αφορούν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις ε, δυνατότητες ε, που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαπιστώσει κατά πόσο είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε κάποια βελτίωση, αλλά τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε στα επόμενα ψηφίσματα για την απαλλαγή να μην είναι υποχρεωμένο το Κοινοβούλιο να κάνει παρατηρήσει επί του θέματο. Αυτέ λοιπόν ω εισαγωγικέ ερωτήσει, βέβαια θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και διμερώ και θα υπάρξουν και άλλοι συνάδελφοι που θα θέσουν ερωτήσει. Ευχαριστώ. Από τους συναδέλφους Κυρία Γκρέσλερ, έχει το λόγο. Πολύ ωραία. Πρώτη φορά νομίζω έχουμε παρόντα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Και είναι η πρώτη φορά νομίζω που μπορεί πέρσι ή πρόπερσι που ασχολήθηκε με θέματα απάτης. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η πρόπερση που ασχοληθηκε με θεματα Καλό λοιπόν θα ήταν να δούμε πόσες περιπτώσεις απάτης έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Χρόνια πόσες περιπτώσεις απάτης έχουν διαπιστωθεί. Και καλό θα ήταν να είχαμε μια εικόνα και του γιατί δεν είχε ενδιαφερθεί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τι μπορεί να κάνει από εδώ και μπρος. Η όλα φυσικά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν μπορεί να ανατρέψει τόσες παγιωμένες πρακτικές και ίσως ε, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αλλάξει πρακτική και να μας πείσει ότι έχει αλλάξει νοοτροπία. Θα ήθελα λοιπόν ε, μια ερώτηση στη συνέχεια, αλλά απευθύνεται στην Επιτροπή και δεν μπορώ να την υποβάλω τώρα. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια ερώτηση ε, στον Επίτροπο Πίμπαλξ, όπου η απάντηση που μου δόθηκε αναφερόταν στο 2008. 84 εκατομμύρια ευρώ νομίζω ήταν η απάντηση ότι χορηγήθηκαν. για 997 άτομα που προσελήφθησαν. 997 άτομα για την περίοδο 2009 με 2011 είναι η περίοδος προσλήψης αυτών των ατόμων. Και αν αυτό αληθεύει, αν όντω προσελήφθησαν περίπου χίλια άτομα για δύο χρόνια, ποιο έλεγε την απόφαση. Εμεί δεν περιμέναμε τέτοιο πράγμα. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάποια δουλειά αναπτυξιακή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αλλά όχι στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί να χρειάζεται χιλιάτομα στις Βρυξέλλες. Ας κοιτάξει λοιπόν η Επιτροπή ε, πώς είναι δυνατόν να μας λέει ε, ότι δεν είναι σε θέση να προσλάβει ούτε ένα νέο υπάλληλο και ξαφνικά να προσλαμβάνει χίλιους από το παράθυρο. Και επιπλέον έχουμε και το ζήτημα των ε, εσόδων από τόκους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με χρήματα ε, σχεδίων. Δεν τους ανήκουν τα χρήματα αυτά. Είναι χρήματα από προγράμματα και σχέδια. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά. Ο Πρόεδρος. Έχουμε τη διαδικασία στον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη τη Απαλλαγή. Ζητήσαμε την Κοκομπίου να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά την εντολή που έχει η τράπεζα αυτή όσον αφορά αυτή συγκεκριμένη αυτή ε, περίπτωση. Η σημερινή συνεδρία συνδέεται συγκεκριμένα με την απαλλαγή. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει και να διαβιβάσει ενδεχομένως κάποια απάντηση. Κυρία Ρολμάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ θερμά. Μια σύντομη επικριτική παρατήρηση καταρχάς. Θα ήθελα την επόμενη φορά να ενημερώνονται και οι συνεισηγητέ ότι υπάρχουν ερωτηματολόγια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Φερρυπίν γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία ούτε τις δικές μας προτάσεις ε, για ερωτήσεις να υποβάλουμε μόνο να δούμε ε, όταν ήταν τελεσμένη η διαδικασία της απαντήσεις. Μια καλύτερη προσπάθεια λοιπόν συντονισμού μεταξύ των συντονιστών. Και προχωρώ στο ερώτημα που ήθελα να υποβάλω. Το εξή λοιπόν, το οποίο επέπεσε στην αντίληψή μου. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταθέτει συνήθω τα χρήματα σε τράπεζες στις εκάστοτε περιφέρειες ή σε ταμεία των κράτων μελών. Σε ποιο βαθμό είναι εξασφαλισμένο ότι θα επιτυγχάνονται και οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών και σε ποιο βαθμό επαληθεύεται πως και τα σχέδια αυτά προχωρούν με βάση τους στόχους και τη στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα όσα έχουμε εμείς προβλέψει. Σε ποιο βαθμό δηλαδή οι στόχοι και η στόχευση επαληθεύονται Υπάρχουν όντως ε, τα σχέδια αυτά, εκτελούνται όπως έχει οριστεί ο στόχος τους, ε, ε, εκτελούνται με στόχο την ανάπτυξη υποδομών, υπάρχει σχετική επαλήθευση και ο συσχετισμός τους με λοιπά συναφή σχέδια, ποιο είναι, γιατί βλέπουμε ότι αναπτύσσονται μερικέ φορέ σχέδια, ένα σχέδιο μεμονωμένο σε κάποιο σημείο απομονωμένο τη Αφρική και τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται για να φέρει καρπού στο σχέδιο δεν υπάρχουν. Επίση, υπάρχουν ε, παληθεύσει και έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην αναπτύσσουν στον ίδιο χώρο δύο-τρία διαφορετικά σχέδια χωρί συντονισμό. Ο συντονισμό δηλαδή μεταξύ των σχεδίων αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνων της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων υπάρχει, λειτουργεί. Επίσης θα ήθελα να δω ένα πλήρη κατάλογο ε, σχεδίων που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πλήρη κατάλογο, εξαντλητικό, όχι αυτό που λέμε highlights of projects, δηλαδή ε, ορισμένα σχέδια ενδεικτικά, γιατί βέβαια είναι εύκολο ενδεικτικά να βρούμε τα καλύτερα και πιο επιτυχημένα σχέδια και θα βγάλουμε από τα ενδεικτικά τον κατάλογο των ενδεικτικών εκείνα τα οποία έχουν αποτύχει, έχουν ε, εμφανίσει καταχρήσεις, διασπάθηση χρημάτων και το καθεξής. Θέλω λοιπόν να ξέρω πόσα σχέδια, σε γιατί ποσό διατίθεται για πόσα σχέδια και για τι ποσό δίδεται η ανάθεση μέσω των ε, δημόσιων προκηρύξεων και βεβαίως πόσες πιστώσεις και εγγυήσεις προσπαθείτε να εξασφαλίσετε. Σας ευχαριστώ, ο κ. Κάφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μάζω έκθεση για την εντολή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα περισσότερα θέματα καλύπτονται. Δεν έχω πολλέ ερωτήσει να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σχολούμαι το θέμα μήνε. Και είμαι στο τελευταίο στάδιο των θεμάτων που συζητούμε. Είναι σημαντικά τα ερωτήματα που ετέθησαν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα χαιρόμουν αν υιοθετήσει σύντομα το Κοινοβούλιο την παράταση της εξωτερικής εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εκεί προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, πώς θα εκτελούνται τα προγράμματα, αυτό που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι, αύξηση της διαφάνειας, μεγαλύτερες απαιτήσει και προδιαγραφές για να εμπλέκονται οι διάφοροι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς όταν είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα αποτελέσματα πρέπει να με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσης συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής τέτοια και θα πρέπει να ταιριάζουν οι στόχοι με τους στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να καταλάβουμε όταν κινούμεθα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε πολύ φτωχές χώρες υπάρχει συγκεκριμένο περιβάλλον εκεί. Δεν προσπαθούμε να βρούμε ε, δικαιολογίες για κακή χρήση πόρων αλλά πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι η ανταγωνιστικότητα σε αυτές τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Διότι όλες οι απαιτήσει για τους φορολογικούς παραδείσους, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τις, στους σκληρότερους κανόνες όσον αφορά την αποφυγή της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Όταν μιλάμε για εκτεταμένη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για περισσότερε πληροφορίε που θα παρέχονται προ το κοινό κλπ. θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τότε γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική από του άλλου, κυρίω όταν κινείται επί εμπορική βάσεω. Ενδιαφερόμαστε όσον αφορά του πόρου Ευρωπαϊκή Ενώση όπω το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και του ίδιου πόρου Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι εμπορική φύσεω. Θέλουμε αυτού να χρησιμοποιήσουμε ή διαφορετικές πολιτικές. Χρειαζόμαστε μια μορφή προσέγγιση πιστεύω. Αναμειγνύοντας χρήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με εμπορικά χρήματα της τραπέζης θα πρέπει να σκεφτούμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτευχθούν αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας με τις χώρες αυτές και να αναγνωρίσουμε τι περιορισμούς θέτουμε σε αυτές τις χώρες και ποιες είναι οι πολιτικοί, ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τι συνέπειες έχει απέτησή μας για διαφάνεια. Με τα χαρά να συνεχίσουμε τη συζήτηση και ελπίζω ότι θα δούμε περισσότερες από αυτές τις ανησυχίες που εκφράστησαν να καλύπτονται από την εξωτερική εντολή που θα δοθεί στην τράπεζα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κανένας βουλευτής δεν επιθυμεί να πάρει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Κίνς, που είναι διευθυντής, αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει κάτι να μας πει σε σχέση με αυτά που μας ανέφερε η κυρία Γκρέσλε. Θέλετε να πείτε κάτι ή όχι. Θα τα μιλήσετε. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στείλαμε επιστολή. Μετά την ακρόαση του Επιτρόπου Πίμπαλξ εδώ, εδώ και 15 μέρες. Να σε εξηγήσω κάτι. Στην εσωτερική συμφωνία για το τέτοιο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης τα κράτη-μέλη διέθεσαν 430 εκατομμύρια συγκεκριμένα για την υποστήριξη δαπανών, να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το κόστος των αντιπροσωπιών και στελέχωση στην έδρα. Ποιο ενδιαφέρον υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Ποια είναι τα συμφέροντα που καλύπτονται. Τα ποιοι είναι οι τόκοι μάλλον από κάποιε καθέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ποσά είναι χαμηλά, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο νομίζω. Η εσωτερική συμφωνία καθορίζει ότι αυτοί οι τόκοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη δαπανών επίσης και όχι για προγράμματα. Για την κινητοποίηση των πόρων ως ήθιστε για τις αποφάσεις χρηματοδοτήσεως. Παρουσιάζουμε μια πρόταση προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως των κρατών μελών. Πρέπει να τοποθετηθούν θετικά και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση. Και τα 430 εκατομμύρια που ανέφερα, αυτή η πόρη είναι η συνεισφορά για το κόστος για όλη την περίοδο 2008 με 2013 για το Ευρωπαϊκό Ανάπτυξη. Το 2008 ελήφθη απόφαση για την πρώτη περίοδο μέχρι το τέλο του 2011. Μέχρι τέλο ενεστώτο έτου. 181 εκατομμύρια που χρηματοδοτούν 942 θέσεις συμβασιούχων και τοπικών υπαλλήλων και 52 θέσεις εδώ με συμβάσεις κάποιο προσωρινό προσωπικό εμφανίζονται αυτές οι θέσεις στο οργανόγραμμα και προσλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και πληρώνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως οι συμβασιούχοι και το τοπικό προσωπικό και τα χρήματα προέρχονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ο έλεγχος διεξάγεται από το ελεκτικό συνέδριο. Θα θεωρούσε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη μέσα αυτού του κόστου χρηματοδοτεί περίπου 50% του κόστου των αντιπροσωπιών ΑΚΕ είναι σημαντική λοιπόν η συνεισφορά αυτή και δεν πρέπει να το θεωρήσετε ότι είναι συμπληρωματικέ θέσει, επιπλέον θέσει. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει καλυπτόταν το κόστο θέσεων που εκαλύπτονται κατά το παρελθόν μέσω του προπολογισμού. Άρα δεν ήταν σε κάθε περίπτωση συμπληρωματικέ πρόσθετε θέσει. Αλλά το 10ο Ταμείο Ανάπτυξη είχε 50% ε, αύξηση σε σχέση με το 1ο. Χρειάζεται και αύξηση του προσωπικού λοιπόν. Όλα αυτά ελέγχονται, όπως σας προανέφερα, από το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, σύντομα παρακαλώ. Πέραν του ότι έχουμε ε, όλη αυτή την ιστορία εκκρεμή, επανέρχομαι στα τόκους Υπάρχουν, υπάρχει περίπτωση τόκοι, έσοδα από τόκους να χρησιμεύουν για την πληρωμή αμοιβών προσωπικού, μισθών δηλαδή. Είναι δυνατόν χάρη σε τόκους να προσλαμβάνεται προσωπικό. Αυτό είναι τελείως λάθος δημοσιονομικά. Θέλετε να δώσετε μια σύντομη απάντηση. Αυτό λέει η νομική βάση. Πριν από το 10 Ταμείο Ανάπτυξη υπήρχε χρήση των τόκων που μπορούσε χρηματοδοτήσει κανεί προγράμματα στο δέκατο. Τα έχουμε περιορίσει και είπαμε στην εσωτερική συμφωνία που εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη ότι οι τόκοι χρησιμοποιούνται μόνο για υποστήριξη δαπανών. Και αυτό ακριβώ κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή το κάνουμε αυτό σύμφωνα με την νομική βάση. Σε όλα αυτά τα θέματα, σε αυτές τις υποθέσεις, έχουμε μεγάλη περιέργεια. Έχουμε δομές που ξέρουμε ότι είναι διακυβερνητικής ε, φύσεως άλλες κοινοτικές. Πολέμησα τους Ευρωπαϊκή Τράπεζα Απενδύσεων να πληρώνει το τιμή της, ε, το χρημάτων που δίνει για την εξωτερική δράση η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα ξαναρυθμίσουμε όλα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δεν ξέρω αν αφορολόγηση των συναλλαγών θα γίνει για να πληρωθούν τα 100 δις της ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως όλα τα μέσα μας τα ξαναεξετάσουμε. Η κυρία Μπαρτόλτ για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να καλύψω όλα τα βασικά θέματα και μετά χαρά να σας δώσω περαιτέρω πληροφορίες, εάν ζητηθούν. Εν είδη αγωγής. Αποτελέσματα και υποβολή αναφορών είναι σημαντικό. Αυτό που αναφέρατε και οι συνάδελφοί μου κατέβαλαν προσπάθεια για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο να ενημερώνουμε το κοινό και εσά. Και ο πλήρης κατάλογος των προγραμμάτων είναι εκεί, από τη σελίδα 76 και πέρα. Και τονίζουμε και τα πιο προβληματικά προγράμματα. Δείχνουμε και τα κενά και τα καλά και τα κακά. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και είναι από τους τομείς που θέλουμε να προωθήσουμε. Σελίδα 49. Έχουμε ένα καλό παράδειγμα ε, διότι βλέπουμε θέσει απασχόληση που δημιουργούνται βάσει των προγραμμάτων της τηλεπικοινωνίας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα εκεί. Αν έρθω εδώ του χρόνου και δεν υπάρχει βελτίωση, ξέρω ότι μου αξίζουν κάποιε επικρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ερωτήματα για τη διαφάνεια, να σας πω ότι ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων και ήθελα διακαώς να βελτιώσω τη διαφάνεια και είδα κατά τη διάρκεια θητείας μου βελτιώσεις στα πρακτικά πράγματο χάρη των συνεδριάσεών μας. Ε, έχω, ε, προσαρμο, έχω ιστορικό στην ανάπτυξη και τώρα προσαρμόζομαι τώρα στον τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν όμως και θέματα πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται λόγω εμπορευματικής, εμπορικής εμπιστευτικότητας. Και πάνω το καταλάβουμε. Κάτι άλλο που ανέφερε ο κ. Κάλφιν και είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν είναι η έλλειψη διαφάνειας για λόγους εμπορικούς, αλλά λόγω ελλείψης ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει η τράπεζα. Διότι χάσετε πολλή δουλειά να παρακολουθεί κάθε κατανομή μέχρι δικαιούχου που μπορεί να παίρνουν 250 ευρώ, τόσο λίγα χρήματα. Ε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε όμως να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση και να θέσουμε πόρους για μεγαλύτερο έλεγχο, θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα μονάδα ελέγχου και καλό θα ήταν να υπάρχει συμπληρωματικό προσωπικό για να αναλάβει τα καθήκοντα. Και εδώ, σε αυτόν τον τομέα, είναι καλές οι κρίσεις για να μας βοηθήσουν ε, να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος. Όμως οι περισσότερες επικρίσεις απέραν από έλλειψη κατανόησης λειτουργίας τραπεζών. Περισσότερο σε αυτό οφειλόταν παρά σε προβλήματα της διαχείρισής μας. Όσον αφορά την απάτη, υπάρχει διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα. Μέχρι το επίπεδο 5. Εκεί που ένας φορέας μπαίνει μια οργάνωση, μπαίνει σε μαύρο κατάλογο. Και έχει συμβεί αυτό. Και είναι κάτι σπάνιο αυτό. Στα πιο κάτω επίπεδα όμως υπάρχει αυξημένος έλεγχος. Και στα τρία χρόνια που ήμουν στο Δικαιωτό Συμβούλιο είδα ότι αυξήθηκαν και οι πόροι και οι διαδικασίες για την καταπολέμηση των απατών. Αυτό αυξάνει τη δουλειά της υπηρεσίας. Είναι πιο σοβαρές διαδικασίες και πιο επαχθείς. Πρέπει να πετύχουμε σωστή ισορροπία. Και πρέπει και αρμόδιοι φορείς να συμφωνήσουν επί των προτεραιοτήτων όσον αφορά την καταπολέμηση των απατών. Αξιολόγηση ελέγχου ετέθη ερώτημα. Κατά πόσο κρίνουμε ότι συμμορφόμαστε με τους στόχους των προγραμμάτων. Και εδώ έχουμε πολλά επίπεδα. Εξετάστηκε ο μηχανισμός επενδύσεων. Πετύχαμε τους στόχους, λέω με τα χαράς. Σε κάποιους τομείς επιδέχομαστε βελτιώσεις. Υπάρχει έλεγχος όμως από τη στιγμή που πέφτει η υπογραφή και οικονομικός έλεγχος όσον αφορά την εκταμείευση και φυσικός έλεγχος που αυτό αφορούσε η ερώτησή σας. Και αυτό μέχρι το τέλος διαδικασίας, μέχρι ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και συντάσσεται έκθεση για το πρόγραμμα. Αν θέλετε ένα έγγραφο και στοιχεία έχουμε πολλά να σας δώσουμε. Κίνδυνος αλληλεπικαλύψεων. Με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους. Χρειάζεται συντονισμός. Εδώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε πρόοδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Συντονισμός μεταξύ κρατών μελών βελτιώθηκε και των διαφόρων φορέων. Στόχος της αναθεωρήσεως του μηχανισμού επενδύσεων και της εξωτερικής εντολής δανειοδότησης διαπιστώθηκε από τον έλεγχο αυτόν ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικό μου καθήκον είναι αυτό, μάλιστα. Καλύτερο συντονισμό. Μπορούμε να έχουμε προσωπικό που θα βοηθούσε σε συντονισμό αν είχαμε επιτόπου προσωπικό. Και τι άλλοι τρόποι υπάρχουν συντονισμού. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Περισσότερα στο μέλλον του χρόνου. Τέλος. Για τη διαγραφή και απάτες. Σπάνιες περιπτώσεις που διαπίστωσα κάτι θητείο μου. Το τμήμα μου έπρεπε να πληρώνει όταν δεν επιστρεφόταν τα χρήματα. Όταν υπήρχε αδυναμία πληρωμής το διαπίστωνα. Σπάνια γινόταν αυτό και οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους σε κανένα δύο χώρες απάτες. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις τώρα που εξετάζονται και δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, διότι ακολουθούνται ιδέωσες νομικές διαδικασίες που δεν έχουν διεκπαιρωθεί. Άρα δεν ενδείκνεται, δεν είναι σωστό να αναφέρω ονόματα. Τώρα έχει, υπάρχει μια γνωστή απάτη, η CDE, θα την γνωρίζετε, συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εντυπωσιάστηκα από την όλη ανταπόκριση της CD. Όταν λαμβάνονται σωστά μέτρα, υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση. Και γι' αυτό έχουμε κάθε πεποίθηση ότι στο μέλλον δεν ξανασυμβεί αυτό. Θα με ανησυχούσε αν δεν είχαμε διαπιστώσει κάποια προβλήματα. Διότι λειτουργούμε σε τέτοια περιβάλλοντα που δεν υπήρχαν προβλήματα, θα σήμαινε ότι θα ήμασταν απρόσεκτοι. Και δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή. Ελπίζω ότι απάντησα σε κάποιε από τι ερωτήσει σα. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κυρία Γενική Διευθύντρια, ευχαριστώ για την παρουσία σα, την παρέμβασή σα. Ευχαριστώ τον συγγετή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλείνουμε αυτό το τμήμα συνεδριώσεω και διακόπτουμε για ένα τρίλεπτο, ούτω ώστε να δώσω την προεδρία στον συνάδελφο Λοιπόν, συνάδελφοι, είμαστε τώρα στο πρώτο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το πρωί. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΕΚΟΝ, η οποία είναι επί της ουσίας Επιτροπή. Ο συντάκτης είναι ο κύριος Οντή. Έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα. για να ετοιμάσουμε αυτή τη γνωμοδότηση, η οποία θα δοθεί στην ΕΚΟΝ. Η ΕΚΟΝ ε, θα ψηφίσει στις 15 Μαρτίου, επομένως εμείς θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει τη γνωμοδότηση στις 28 Φεβρουαρίου. Να δώσω λοιπόν απευθείας το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Euh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να χαιρετήσω εδώ την παρουσία του κυρίου Ντομίνικ Τεκραϊανκούρ, εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι και των θεσμικών ζητημάτων. Και θα ήθελα να ευχαριστώ και για την ευαισθησία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις θέσεις των βουλευτών. Η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή Στι δύο πρώτε παραγράφου εκφράζει την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να παρακολουθεί την ουσιαστική κίνηση των στρατηγικών επενδύσεων μέσω και μακροπρόθεσμα με βάση της, ε, την εμπειρία που έχουμε συλλέξει. Επίσης, συντασσόμαστε με την άποψη στο σημείο 3 ότι είναι επιτακτική να εκνοητηρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την αξιολόγηση 3α Ω προ την επιστροπτική τη ικανότητα, γιατί άλλωστε την αξίζει. Και αυτό το σημειώνω γιατί εξηγεί και τι θέσει που έχουμε υιοθετήσει στις περαιτέρω ε, παραγράφους. Το λέω διότι πολλέ φορέ σε μέσο και μακροπρόθεσμε επενδύσει ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προβλέπεται πάντα κάτι σαν το Μαϊντανό δηλαδή. Αν όμω συνεχιστεί αυτό και αναλαμβάνει κίνδυνο ο οποίο δεν είναι συμβατό με τι παραδοσιακέ ε, μορφές και τους παραδοσιακούς τύπους πιστώσεων, τότε διατρέχει υπερβολικά υψηλό κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεν έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω, όταν λέει ότι πρέπει να χορηγεί επιδοτήσεις, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Για την Οικονομική Επιτροπή θα ήθελα να υπενθυμίσω, Πρόεδρε, ότι το καταστατικό ορίζει πως εμείς ε, είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας Επιτροπή ε, και κατά προκλειστικότητα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ξέρω ότι ε, γίνεται μια ρύθμιση και το εναλλάσσουμε καθέτος το ποιο θα λάβει την έκθεση, αλλά στον κανονισμό ορίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχει την αρμοδιότητα και πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Παράγραφο 4, με τη σημαντικότερη πρόταση για μένα, και θα ήθελα εδώ απάντηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί δεν έχω καταφέρει, δεν καταφέρνουμε να πείσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ασκεί τον ρυθμιστικό και προληπτικό έλεγχο που οφείλει. Και για να εξηγηθώ, όταν ήμουν εισηγητή, δεν, θυμάμαι, δεν θυμάμαι πια το έτο, είχα συζητήσει μάλιστα με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τον διοικητή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που, ε, τον κύριο Βίδεν, ο οποίο είχε πει ότι συμφωνεί πω θα πρέπει να έχει ρυθμιστικό ρόλο, όπω όλε οι εθνικέ τράπεζε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καθώ όμω είναι διεθνή οργανισμό, όπω η, η Παγκόσμια Τράπεζα και το καθεξή, η ΕΤΕΠ δεν υπάγεται σε ρύθμιση έχει εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου και επιτροπή ελέγχου κτλ. Αλλά δεν έχει πραγματική αποστολή προληπτικού ελέγχου, η οποία θα εξασφάλιζε την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών, τη βέλτιστε εγγυήσει, τη εγγυήσει ιδίων πόρων, ιδιαίτερω έναντι τρίτων. Έτσι λοιπόν αυτό το προληπτικό έλεγχο σκεφτήκαμε να τον εγγράψουμε στο άρθρο 127 τώρα, το με την παλιά συνθήκη, με επί τι το άρθρο, στην έκτη παράγραφο όπου το Συμβούλιο μπορεί ομόφωνα να αναθέσει προληπτικό έλεγχο ως προς την θέσπιση πιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και είχαμε συστήσει το θέμα αυτό με τον κύριο Μέιστατ και είχε συμφωνήσει, όπω είπα. Μόνο το Συμβούλιο δεν συμφώνησε τελικά. Ούτε και η Επιτροπή κατέθεσε αντίστοιχη πρόταση ποτέ. Εγώ έκανα γραπτή αίτηση, γραπτή πρόταση μάλλον προ το Συμβούλιο. Το οποίο μου απάντησε, άμα δεν μου έχει ζητήσει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν Επιτροπή διστάζει να καταθέσει την πρόταση, γιατί ξέρω το Συμβούλιο δεν πρόκειται να συμφωνήσει με πλειοψηφία. Άρα δεν προχωράει η υπόθεση. Και έτσι, με τη θέσπιση τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, κατέθεσα δύο τροπολογίε, τι οποίε έκανε δεκτέ η Οικονομική Επιτροπή, γιατί το είχα συζητήσει με και απερίφθησαν σε επίπεδο τριμερού διαλόγου. Δηλαδή, είχα υπολογίσει αυτή τη ρύθμιση να την εγγράψω μέσα στην Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Και καθώς το καταστατικό της ΕΤΕΠ εξαρτάται από τη συνθήκη, δεν είναι δυνατόν μέσα σε ευρωπαϊκό νομοθέτημα να εισαχθεί τροποποίηση που θα αναιρεί κάποια διάταξη της συνθήκης. Ήταν βέβαια η αντίρρηση μάλλον τυπολατρική κατά την άποψή μου, εγώ πάντως δεν υποχωρώ. Πάντως για λόγους νομικούς φαίνεται ότι τώρα δεν μπορεί να γίνει η ρύθμιση, δεν μπορεί να ε, αναλάβει αυτή την αρχή ή αυτή την, ε, αυτό το προληπτικό έλεγχο μάλλον η τραπεζική αρχή. Ε, γι' αυτό περνώ και στην πέμπτη παράγραφό μου όπου είτε θα επανέλθει αυτός ο ρυθμιστικός έλεγχος βάσει του άρθρου 127 όπου θα επανέλθει η Επιτροπή δηλαδή για να πει ναι αναθετήθεται τώρα πλέον αυτός ο έλεγχος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε η ΕΤΕΠ εθελοντικά προτείνω να υπαχθεί στο προληπτικό έλεγχο μιας αρχής που μπορεί να είναι είτε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είτε μια ανεξάρτητη ελεκτική αρχή. Και το, η προσωπική μου ιδέα είναι η εξής. Ότι εφόσον μπορούμε και θέλουμε με μακροπρόθεσμα να επενδύουμε με τα ευρωομόλογα κλπ. Αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί επισημένω προ την έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το διαβάσει κανεί το κείμενο. Υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των Eurobonds, αυτά που ονομάζω ξεκάθαρα project bonds, δηλαδή ομόλογα που είναι ε, συγκεκριμένα εστιασμένα στην εκτέλεση ενό σχεδίου και τα λοιπά ευρωομόλογα, τα οποία είναι τελείω διαφορετική υπόθεση. Λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε. Εγώ μιλώ τώρα για τα συγκεκριμένα σχέδια υποδομών, ομόλογα για σχέδια υποδομών. Εδώ λοιπόν είναι απαραίτητο και πιστεύω θα πρέπει όλοι μαζί να το αναλογιστούμε, να εξετάσουμε και πάλι την χρηματοδότηση ή μη τι άλλο αυτών των υποδομών και των σχεδίων υποδομών. Γιατί υπάρχει ανάγκη. Μέσα επίσης υπάρχουν, ίσως χρειαστεί όμως να δημιουργηθούν και νέα. Και γι' αυτό αναφέρομαι και συνεχίζω με την παράγραφο 6 στην πρόταση την οποία επαναφέρω από το 2006 που είχε αρχικά υποβληθεί να μπορέσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει στην ΕΤΕΠ μια ευρεία μελέτη του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις γιατί η ΕΤΕΠ έχει προσωπικό εξαιρετικό στο Λουξεμβούργο με γνώσεις από το δημόσιο, τον ιδιωτικό, τον τραπεζικό κλάδο που θα μπορούσαμε λοιπόν να τους αναθέσουμε μια μελέτη για το πώς μπορούν, είτε στις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε σε επίπεδο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, να ε, προσδιορίσουν μέσα χρηματοπιστωτικά για την επένδυση σε μακροχρόνιο επίπεδο αυτών των υποδομών. Μια βάση δηλαδή, όπως προσδιορίζω και στη γνωμοδότησή μου, για πολιτικό δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μετά την πρόταση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Eurobonds. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκτό από την κυρία Γκρέσλε θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, ο κύριος Κάλφιν. Ωραία. Να ακούσουμε καταρχάς ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει ο κύριος Δεκραϊανκούρ και μετά δεν ξέρω αν θέλει να λάβει το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στις δύο βασικές παρατηρήσεις που γίνονται στη γνωμοδότηση του κυρίου Ντί. Η πρώτη αφορά την εποπτεία και η δεύτερη ε, μία μελέτη για τη χρηματοδότηση. Για το θέμα της εποπτείας, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε με τον εισηγητή και συμφωνούμε εδώ και χρόνια. Η τράπεζα είναι διατεθειμένη να δεχτεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη μορφή εποπτείας, εάν, και αυτό το εάν είναι σημαντικό, ε, μπορεί να το επιτρέψει αυτό ο κανονισμός και τα όσα γράφουν οι συνθήκες. Καταρχάς, κανένα από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν αποτελεί αντικείμενο εποπτείας και δεύτερον, κανένας δεν έχει την εποπτεία που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα επανέλθω από αυτού. Και τρίτον, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι εθνικοί ε, επενδυτές που κάνουν αντίστοιχη δουλειά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως δεν αποτελούν αντικείμενο εποπτείας. Και η εποπτεία είναι κυρίως θέμα της προστασίας των καταθετών και δραστηριότητες ε, των ε, τραπεζών, δραστηριότητες που δεν διεξάδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επιδίσεων ή οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες ανάλογης ε, φύσεως. Και αυτός είναι και ο μόνος λόγος για τον οποίο ε, θεωρούμε ότι είμαστε συγκρίσιμοι με όλους τους ομόλογούς μας. Οι θέσεις μας δεν είναι ακόμα ισχυρότεροι διότι η συνθήκη και το κανονισμό της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων ε, προβλέπει να έχουμε μία ανεξάρτητη επιτροπή εποπτείας. Κάτι το οποίο δεν έχει κανένας άλλος από τους ομολόγους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Ενισχύεται δε από τη συνθήκη της Λισαβόνας διότι υπάρχουν επιπλέον μέλη τα οποία θα πρέπει να ε, έχουν και υπόβαθρο εποπτείας και έχουμε ανθρώπους ε, οι οποίοι φυσικά βασίζονται και σε εξωτερικούς ε, ελεγκτές. Υπάρχει λοιπόν μια εσωτερική δομή η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι και ισχυρότερη από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα με την οποία μπορούμε να συγκριθούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είμαστε διατεθειμένοι και όπω πολύ σωστά όμω εξήγησε ο εισηγητή σα, υπάρχει δυσκολία διότι δεν υπάρχει απαιτούμενη ομοφωνία για να ε, διεξάγει αυτά τα καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα ήταν και πιο λογική προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικέ λύσει. Ε, κατόπιν δική σα προτάσεων συζητήσαμε με την ε, νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αλλά υπάρχει και το νομικό πρόσκομα που αναφέρατε εσείς, αλλά υπάρχει και το θέμα των δυνατοτήτων τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν τους ελέγχους. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι, ε, και αυτό ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια, να έχουμε ένα πολύ στενό διάλογο και συνεργασία με την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου και χάρη σε αυτόν έχουμε ένα πολύ ισχυρό επιπλέον εποπτικό στοιχείο διότι ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης μπορούσαμε να είχαμε επαναχρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η επαναχρηματοδότηση βέβαια σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται τα οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται μέσω της αρχής του Λουξεμβούργου. Ε, πρόκειται για ένα περαιτέρω βήμα το οποίο νομίζω συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις. Ε, αυτό το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα στο κείμενο είναι η ιδέα να υπάρχει και ένας ακόμα εξωτερικός ανεξάρτητος ε, επόπτης. Το έχουμε ήδη έναν και το να έχουμε και άλλους τρεις-τέσσερις δεν θεωρούμε ότι είναι και ιδανική λύση. Ε, οι άλλε δύο εναλλακτικέ λύσεις, είτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, κατά αν αυτό είναι πολιτικό δυνατόν, ή η ενίσχυση του έργου μας με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και έναν εθνικό επόπτη, θεωρούμε ότι είναι η καταλληλότερη λύση. Για το θέμα τώρα της μελέτης που προτείνεται για να εξετάσει νέους τρόπους ε, χρηματοδότησης ε, κυρίως υποδομών θεωρούμε ότι είναι εφικτό. Γίνεται αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας πω, διότι αυτό που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανάλυση που γίνεται αυτή τη στιγμή ως προς τη δυνατότητα να έχουμε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές λίγο πολύ καλύπτουν τις απαιτήσει αυτής της μελέτης, τις οποίες θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε, να τις επισημοποιήσουμε και να τις ε, διαμορφώσουμε βάσει των απαιτήσεών σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το θέμα του ανεξάρτητου τμήματος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Βέβαια αυτό μάλλον δεν είναι θέμα της τράπεζας, είναι μάλλον θέμα της Κομισιόν. Ε, τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, ε, συμφωνώ για την παρατηρήση σας για τα ομόλογα, τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Ε, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τα οποία υφέρπουν πίσω από αυτή τη διατύπωση. Η χρήση του όρου είναι ατυχή Να σας πω ότι τα ομόλογα τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεις είναι ευρωπαϊκά ομόλογα, δεν είναι τίποτα άλλο. Και κάθε χρόνο κυμαίνονται στα 60 δις ανά χρόνο για να ε, χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της τράπεζας. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πρόταση του ε, κυρίου Μπαρόζο να έχει τα project bonds, αυτά τα ομόλογα, τα οποία να σας πω ότι δεν είναι ευρωπαϊκά ομόλογα, είναι ομόλογα τα οποία θα εκδίδονται από όσους προάγουν επενδυτικά προγράμματα, από τον ιδιωτικό τομέα δηλαδή. Δεν ε, δημιουργούν καμία δέσμευση ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτε για τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να καλούνται λοιπόν ευρωπαϊκά ομόλογα, αλλά project bonds. Και υπάρχουν και αυτή την ιδέα για τα ομόλογα για το ε, δημόσιο χρέο ή τη ενίσχυση του προπολογισμού που είχε ο Ντελόρ τότε. Με συγχωρείτε που τα αποκαλώ ομόλογα Ντελόρ, Γιούγκερ ή Μπαρόζο. Πρόκειται για τελείω διαφορετικά ομόλογα. Τα ομόλογα Μπαρόζο λοιπόν δεν δεσμεύουν τα κράτη-μέλη ούτε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Καζόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επικεντρωθώ σε αυτά τα δύο σημεία. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Ντί διότι συνόψισε επακριβώς την κατάσταση για το θέμα της ε, δημοσιονομικής εποπτείας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εμεί συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για το πόσο θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να διασφαλίσουμε ότι θα έχει την ίδια άριστη ε, την περιφορά που έχει τώρα. Υπάρχουν βέβαια και θέματα ε, που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή, Τράπεζα, ε, συγγνώμη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και το κατά πόσον μπορούν αυτές να ασκούν το ρόλο του επόπτη. Η τρίτη ιδέα που προτείνεται το να γίνουν κάποιες ε, άτυπε διευθετήσει με άλλου φορεί και εδώ να πω ότι καταλαβαίνω ότι το να υπάρχει μία επιπλέον εξωτερική αρχή εποπτείας να μην προσθέσουμε ένα επιπλέον επίπεδο, αλλά να έχουμε έναν εθνικό επόπτη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να εξετάσουμε δηλαδή αυτά τα ενδεχόμενα περαιτέρω και όχι κάποιους έξτρα επόπτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό για τις επόμενες πολιετήσεις δημοσιονομικές προπτικές Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Τράπεζας Επενδύσεων που διευκρίνησε ότι πρέπει να ρίξουμε λίγο φως ε, περαιτέρω για τα ομόλογα. Ε, τι είναι τα project bonds που προτείνει ο κύριος Μπαρόζο, πρέπει να τα δούμε λίγο ε, πιο αναλυτικά. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα να έχουμε ιδιωτική χρηματοδότηση για σημαντικά προγράμματα και ε, επειδή προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, πρότασή της για τις επόμενες δημοσιονομικές ε, προοπτικές, ετοιμάζουμε, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μία ανάλυση για να διασφαλίσουμε ότι η σωστή χρήση αυτών των νέων μέσων θα μας βοηθήσει και ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διότι έχει και την ανάλογη εμπειρογνωμοσύνη για το πώς λειτουργεί η αγορά που μας βοηθά. Όπως σας είπα, η ανάλυση αυτή γίνεται στα πλαίσια της προετοιμασίας των νέων δημοσιονομικών προοπτικών να σταθώ και στο θέμα των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Είναι πολύ σημαντικό και για σας. Το είπα και προηγουμένως στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ε, καθορίζει Ε, κάπως και το τι γίνεται με το Κοινοβούλιο. Εάν αυξάνονται αυτά τα μέσα θα πρέπει να αυξηθεί και ο έλεγχος από πλευράς ε, ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να έχουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και κανόνες ώστε να υπάρχει και μια σαφής διάφανη έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να μπορούν να ελέγξουν καταλήλως την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καζόλη. Τέσσερις παρεμβάσεις έχουμε επιπλέον. Και μετά, επειδή πρέπει να συζητήσουμε και την απαλλογή προ του Οργανισμού, θα πρέπει να είμαι πολύ αυστηρό, Δύο λεπτά ο καθένα. Η κυρία Γκλέρ. 19,2 e δισεκατομμύρια ευρώ είμαστε ε, μέσω προς τον, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τη σχετική ευθύνη και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι εδώ και η υποχρέωση λογοδοσίας και η ευθύνη η πραγματική υπάρχουν και δεν βλέπω ακόμη να έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα. Γι' αυτό θα πρέπει θέλω να καταθέσω άλλε τροπολογίε. Προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ήθελα να ρωτήσω τι εννοεί ω subsidiaries. Σημαίνει θηγατρικέ, όπω έχω δει μερικέ φορέ να μεταφράζεται, ή κάτι άλλο. Γιατί βέβαια εδώ μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέτει, να αναθέτει περαιτέρω καθήκοντα στην ΕΤΕΠ και κομμάτια ολόκληρο του προπολογισμού για διαχείριση. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό στο μέλλον και σε ποιο βαθμό θα αναλαμβάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τέτοιου είδους καθήκοντα. Επίσης θα ήθελα να μάθω τι εννοεί ω δημοσιονομικά μέσα. Και μια και είμαστε εδώ έτσι όλοι μια όμορφη παρέα, μπορείτε να μου εξηγήσετε και αυτό. Τι σημαίνουν δημοσιονομικά μέσα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκάι τις στο λόγο. Αλλά δεν θα τον λάβει, θα μιλήσει η κυρία Χέρτσοκ εκ μέρους ομάδας του. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια του κυρίου Ντί και ήμουνα και στην άλλη επιτροπή, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, όπου εκεί είδαμε ότι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες της είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και πετυχαίνουν τους στόχους. Συμφωνώ απόλυτα αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να διαθέσουμε περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα μέσα του συστήματο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λειτουργεί σωστά και ότι αυξάνεται η διαφάνεια και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εποπτείας. Καλωσορίζουμε την ιδέα του κυρίου Ντί, του εισηγητή, που ακολουθεί την κατεύθυνση, ο ρυθμιστικός έλεγχος θα πρέπει να η χώρα, Όμω έχουμε διαφορετική άποψη περί της ρυθμιστικής αυτή εποπτείας ο κ. Σοντή πρότεινε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. διότι δεν είναι θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δέκα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Πώς μπορούν να υποπτεύουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αν δεν είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενδιαφέρουσα ιδέα μεν, πρόβλημα δε, διότι βάσει των συνθήκων δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η εποπτεία. Εν τί αυτή περιπτώση πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα. Η άλλη ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σαν ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας μπορεί να κινηθεί σε αυτό το επίπεδο. Ε, ενδιαφέρον αυτό, αλλά δεν είναι εποπτικό όργανο. Σημαντικότατο ζήτημα. Χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Ενδελεχέστερη ανάλυση. Θα ήταν σημαντικό η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βρει μια διέξοδο. Υπάρχει θέμα προς επίλυση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι για την επίλυση όμως. Ίσως οι τραπεζικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αλλάσσονται κυκλικά. Δεν ξέρω. Συμφωνούμε το στόχο, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε. Ας το εξετάσει λοιπόν περαιτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρει την ενδεδειγμένη λύση. Η οποία τελικά θα πετύχει τον ευκταίο στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος θα πρέπει να γίνει προβληματισμός, συζήτηση μεταξύ της ομάδας Σενδί και του Σικτυκίου Χατζημαρχάκης. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η Χέρτσοκ, γιατί δεν είμαι και εγώ πεπισμένο ότι είναι καταλληλότερο χώρο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά, εν πάση έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική τώρα, την οποία έχουμε και εμεί προαγάγει ω Ευρωβουλευτέ, την ε, τραπεζική εποπτεία δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι ήδη έγινε μια παραπομπή στην, Ευρωπαϊ... στην Λουξεμβούργιανή εποπτική αρχή από τον ομιλητή νωρίτερα. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο κείμενο, θα πρέπει να ε, ξεκαθαριστεί αυτό και ίσως να είναι σκόπιμο να βρει η κάθε μία από αυτές τις εποπτικές αρχές τον κατάλογο συνομιλητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι πριν από καμιά δεκαετία μέρες περίπου έγινε μια ακρόαση στην πολιτική μου ομάδα ε, για το θέμα της χρηματοδότηση στο μέλλον και βέβαια τα Eurobonds ε, είχαν προέχουσα θέση στην υπόθεση αυτή και πολύ καλή υποδοχή. Πρώτα απ' όλα βέβαια πρέπει να πάντοτε να γίνεται η διάκριση των διαφόρων ειδών ομολόγων για να μην μπαίνουν όλα μέσα στο ίδιο καλάθι. Σε ορισμένε χώρε τα ευρωομόλογα είναι ε, λέξη Κακοί, δηλητηριασμένοι θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, θα πρέπει να συστήσουμε τις προτάσεις, είτε είναι του Juncker είτε οποιοδήποτε άλλου. Και βέβαια στην Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό των ομολόγων, διότι κύριε Κρένκορ δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς παρόν εκεί σε μια προηγούμενη συνεδρίαση για την απαλλαγή, όπου είχαμε επισημάνει τις ε, ελλείψει σε επίπεδο επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα ω προ την αξιοποίηση των κονδυλίων. Δεν είμαστε θέση δηλαδή να προσφέρουμε τη λεγόμενη προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία σε τέτοιου είδου μεγάλα σχέδια. Τα σχέδια όμω τα οποία χρηματοδοτεί η δική σα τράπεζα την καταφέρνουν αυτή, την εξασφαλίσουν αυτή την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει στην, στην Επιτροπή μα Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Δηλαδή, πρέπει πάντα να πρόκειται για δωρεέ grant, δηλαδή χρήματα που δώριζουμε, που χαρίζουμε, ή θα μπορούσε να είναι δάνειο με προς την τις τη επιστροφή των χρημάτων, ώστε να γίνει μια δουλειά, μια επένδυση. Ή μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεικτή, ε, να βρούμε μια μεικτή λύση, δηλαδή να αναμίξουμε τη δωρεά με το δάνειο, το grant με το loan. Και από τα έχω ακούσει, αυτά που έχουν σαν πολύ καλό αποτέλεσμα τα risk shared finance facility, δηλαδή μέσα χρηματοδότησης με καταμερισμό κινδύνου είναι μέσα τα οποία δεν είναι καινούρια, δεν είναι καινοφανή, υπάρχουν στην αγορά εδώ και χρόνια, δεν τα γνωρίζουμε εμεί αρκετά καλά και δεν τα έχουμε αξιοποιήσει αρκετά, αλλά εξασφαλίζουν πολύ περισσότερη αποτελεσματικότητα και θα πρέπει νομίζω να τα συστήσουμε πιο προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκάλφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι εν γέννη συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του Ζαν Πιέροντι σχετικά με την έκθεση. Κάποιες σκέψεις έχω όσον αφορά την εποπτεία και τη ρύθμιση. Χρειάζεται η εποπτεία όταν υπάρχει συστημικός κίνδυνος κανονικά. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διατρέχει συστημικό κίνδυνο. Οπότε θα πρέπει να δημιουργηθεί εποπτικό φορέας που το διορθώνει αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια. Όμω, πρέπει να συγκρίνουμε τους κανόνες για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνάρτηση με άλλου ευρωπαϊκούς επενδυτικούς φορείς. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ίσω θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Αυτό προτείνατε να υπάρχει κάποια θελοντική παρουσίαση πληροφοριών κλπ. κλπ. Αυτό ίσως να είναι ε, κάτι θετικό. Εν συγκρίση βέβαια με άλλους ανάλογους διεθνείς φορείς. Ο συστημικός κίνδυνος όμως δεν πρέπει να συνδέεται σαν έννοια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν θέλουμε να ασχοληθούμε με τους διεθνείς χρηματοστητικούς οργανισμούς, από αυτή την έποψη θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Επίση, είναι πολύ καλή ιδέα να έχουμε την άφηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και θα ήθελα να επενθυμίσω ότι με την οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εφήβρε νέα μέσα, νέα εργαλεία. Πρότεινε τέτοια εργαλεία και ήταν πολύ επιτυχή, ακολουθώντα τι προτεραιότητε που ετέθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμω ότι όταν αναφερόμαστε στι επενδύσει και τι προοπτικέ για αυτέ, καταρχά θα θέλαμε να δούμε ποιε είναι οι δημοσιονομικέ προοπτικέ που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται ότι θα παρουσιαστούν τα μέσα ενστότοσέ έτους για να δούμε ποιε θα είναι οι προτεραιότητε των επενδύσεων. Ε, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο των επενδύσεων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα πρέπει εκεί να εντάξουμε τις δυνατότητες που θα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δυνατότητες για να συμβάλλει στις επενδύσεις ε, με διάφορα ομόλογα για συγκεκριμένα προγράμματα κλπ. Project bonds ή άλλα μέσα. Και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να παράσχει ε, διάφορε γνώσει. τεχνογνωσία. Οι προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωση που να καθοριστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να δω πώ αυτέ θα αντικατοπτριστούν στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οι απαντήσει ο κ. Στεκάκο, θέλετε να απαντήσετε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που υπόθηκαν. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλώ λέει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Και Κύριε Κασόνη. Λοιπόν, για να κλείσει ο εισηγητής, ευχαριστώ. Καταρχάς όσον αφορά τη ρύθμιση, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ ελέγχου ότι τα από τη ρύθμιση δεν έχουν σχέση. Ένας ελεγκτής κάνει μια δουλειά είναι κάτι ξεχωριστό. Η ρύθμιση αυτή γίνεται από δημόσιο φορέα που αφορά τη ρύθμιση των χρηματιστικών οργανισμών σε όλα τα κράτη-μέλη και εμεί ψηφίσαμε μια Ευρωπαϊκή Αρχή ρύθμιση. ρύθμισης. Δεν έχει σχέση με τον έλεγχο. Αν εγώ αναφέρθηκα στον ανεξάρτητο ελεγκτή σαν ιδέα, διότι εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθώ να βρω μια δημόσια λύση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια λύση, διαρωτήθηκα μήπω εθελοντικά θα μπορούσαμε να αναθέσουμε μια υπεργολαβία σε φορεί ιδιωτικού. Αλλά είναι η τελευταία λύση, έσχατη λύση, διότι δεν μπορώ να βρω λύση. Ευχαριστώ κυρία Χέρτσογκ που προτείνατε να μας διαφωτίσει από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω το εξή. Εφόσον δεν βρίσκουμε λύση, ε, θα θεωρηθεί ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Το λέω φιλικά προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εκτιμώ αφάνταστα. Βλέπω ποια είναι η απάντηση, μου λένε συμφωνώ, συμφωνώ. Και κάθε φορά δεν βρίσκουμε λύση. Δεν πρόκειται περί πονιών. Ξέρω ότι υπάρχει διαφάνεια, βούληση κλπ. Ότι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχουν υπάλληλοι πολύ ποιοτικοί κλπ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ρύθμισης γενικό. Τα, οι αρχηγοί κατών και οι κυβερνήσεων Μα είπαν στην αρχή. Μετά από την κρίση κανένα μέσο, καμία δομή, κανένα φορέα δεν θα κινείται χωρίς ρύθμιση. Και στο ημικύκλιο υπήρχε και αυτό. Ο Μισελ Μπαρνιέ μας είπε σε ένα συμπόσιο και μας είπε δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν ούτε ευκταίο να προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τις τράπεζες, τις δημόσιες, για την ανάπτυξη. Διότι, λέει ο Μπαρνιέ, κανένας δεν θα είναι άνευ ρύθμισης. Μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει ρύθμιση και κανείς δεν το λέει και εδώ και τέσσερα χρόνια δεν βρίσκουμε λύση. Συμφωνώ με όλες τις λύσεις. Μπορώ να πω σε τροπολογίες μας και να πω να αναθέσουμε μια μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Το να αναθέσουμε στην αρχή της, ε, του Λουξεμβούργου, να εμπιστευτούμε την αρχή της Λουξεμβούργου. Θεώρησα όταν είδα τις προδιαγραφές και την εντολή, είπα ότι είναι ατελής και ότι ήθελαν κάποιες συμπληρώσεις. Το Λουξεμβούργο είναι μια χώρα που έχει πολλές τράπεζες, ως αφορά το Τραπεζών, ε, δεν θα κρίνω ποια είναι η άποψη που έχει ο κόσμο όσον αφορά τον έλεγχο που διενεργεί το Λουξεμβούργο επί των τραπεζικών των οργανισμών. Λοιπόν, ας, ας υπάρχει κυκλική εναλλαγή ίσω των ελεκτικών φορέων και μπορούν να συντονίζονται εντό τη δομή τη συντονιστική, δεν ξέρω πώ πώς καλείται, που εδρεύει στο Λονδίνο. Γιατί να μην έχουμε την αρχή του Λουξεμβούργου να υπάρχει ένας κανονισμός που θα λέει ότι οι αρχές του Λουξεμβούργου θα, κάνουν αυτό, θα εκτελούν αυτό το σκοπό του ελέγχου. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Για την άλλη ιδέα, να μην υπάρχει ρύθμιση, έλεγχος, ε, ε, αυτό σίγουρα δεν είναι επιχείρημα. τα κεφάλαια προέρχονται τα κράτη-μέλη. 260 εκατομμύρια από τις συνθήκες. Τα κράτη-μέλη δώσαν ε, τελικά ελάχιστα. Και έχετε το τριπλό α λόγω των εγγύσεων της συνθήκης. Και είναι δημόσια χρήματα, δεν είναι καταθέτες. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις διότι είσαστε υπερεθνικός φορέας. Και δεν υπάρχει υπερεθνικό όργανο ούτε η Παγκόσμια Τράπεζα ούτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει υπερεθνικό φορέα που έχει έλεγχο. Εάν το κάνουμε εμεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δώσουμε το παράδειγμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ένα μέρο του κόσμου που δίνει παράδειγμα, ε, ακολουθεί την ευρωπαϊκή παράδοση. Ευχαριστώ του συναδέλφου που στηρίζουν την ιδέα τη μελέτη, διότι στα ευρωομόλογα δεν βγάζουμε άκρη. Θέλουμε μια μελέτη ποιότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε με του φορεί ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα, όσον αφορά τι μακροπρόθεσμε επενδύσει, θα μα εξυπηρετούσε όσον αφορά τι τροπολογίε, όσον αφορά τι εγγύσει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν την υπέβαλα, διότι όπω όλοι οι βουλευτέ, περίμενα τι τροπολογίε για να μπορέσω και εγώ να τροποποιήσω αναλόγω και να ελέγξω το μέγεθο τη εκθέσεω. Ευχαριστώ κύριε Οντή, λέει ο πρόεδρο. Έχουμε γνωμοδότηση λοιπόν. Οι τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι και μετά θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση 28 Φεβρουαρίου. Θα υπάρξουν πολλές διμερείς επαφές και θα μπορείτε να έρθετε σε επαφή και την, με τους κοιόδης ηγητές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φτάνουν στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας. Η απαλλαγή προς τις διάφορες υπηρεσίες. Ο κ. Σταυρακάκης είναι ο εισηγητής μας. Έχουμε 50 λεπτά στη διάθεσή μας. Αρχική εισαγωγή από τον κύριο Οσί από το Ελεκτικό Συνέδριο. Μπορείτε να μας κάνετε μια εισαγωγή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Προτείνω να δούμε σήμερα δύο οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Στήμα και το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ήρθαμε εδώ σήμερα, κύριε Πρόεδρε, για να δώσουμε κάποια στοιχεία και σε εσά και στους συναδέλφους. Καταρχάς για το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Σώμα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό συζητήθηκε εχθές ε, για τα θέματα της απολογής για το 2009 και θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, έχω να σας ε, περιγράψω μια ιστορία για τον έλεγχο του 2009. Όταν ξεκινήσαμε να διεξάγουμε τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι είχαμε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία των προσωρινών λογαριασμών για το 2009. Λογικά μεν, γιατί δεν υπήρχε εξειδικευμένος λογιστής ε, στον οργανισμό και υπήρχε μία ε, καθυστέρηση ε, λογαριασμών ενός ε, εκατομμυρίου ευρώ τα οποία δεν είχαν εισαχθεί στον έλεγχο κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση ήταν χαόδης. Το ε, θέμα διευθετήθηκε σε τρεις αποστολές για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο. Όλα άλλαξαν βέβαια όταν προσελήφθη νέος ε, διευθυντής ε, και νέος επικεφαλής διοίκησης. Προσελήφθηκε προσωρινά ένας λογιστής από μια λογιστική εταιρεία για να εξεγετάσει τα θέματα και ε, οι λογαριασμοί για το 2009 εγκρίθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, υπάρχει όμως και ένα σημείο με τον οποίο αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στις αρχές του 2009 για την προετοιμασία των λογαριασμών. Ε, οι λογαριασμοί είναι εγκεκριμένοι για το 2009, ε, θεωρούνται ότι είναι ε, εντάξει. Βρήκαμε κάποια προβλήματα με τις προμήθειες. Θεωρήσαμε ότι οι διαδικασίες προμηθειών και οι κατάλληλοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί δεν ακολουθήθηκαν από τον οργανισμό. Και επίσης διαπιστώσαμε ότι για την πρόσληψη συμβούλων και εκπαιδευτικών επιρρογνωμόνων η διαδικασία ε, δεν έγινε μέσω διαγωνισμού. Επίσης υπήρχαν κάποια θέματα προσλήψεων και θέματα που σχετίζονται με τις ταξιδιωτικές δαπάνες. Εχθές ο διευθυντής του οργανισμού μας ανέφερε ότι πολλά από αυτά τα θέματα ε, πλέον ε, αντιμετωπίζονται και έχει γίνει εισαγωγή ενός ε, προγράμματος διαχείρισης, κάτι το οποίο ζητήσατε εσείς ε, κύριε Πρόεδρε και οι συνάδελφοί σας από πλευράς Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Αυτά ως εισαγωγικά σχόλια. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, τουλάχιστον για το οργανισμό της αστυνομίας ε, και στους επόμενους ελέγχους, αλλά αυτό βέβαια ε, Να περάσω τώρα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Κύριε Πρόεδρε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων εδρεύει στο Λονδίνο. Δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό. Έχει ε, προσωπικό 6.064 άτομα, τουλάχιστον για το τέλο του 2009 και είχε έναν ε, προπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πολύ σκληρή δουλειά, δίνει άδεια για φάρμακα, για ανθρώπινη χρήση αλλά και για κτηνιατρικά φάρμακα για του κατοίκου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα να κάνω αρκετά σχόλια και θετικά αλλά και αρνητικά. Να χρησιμοποιήσω τη Mary Poppins. A spoonful of sugar would help the medicine go down. Μια κουταλιά ζάχαρη θα βοηθήσει το φάρμακο να το καταπιείτε καλύτερα. Το ελεγκτικό συνάδελφο θεωρεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων λειτουργεί καλά. Ε, έχω, δεν υπάρχει θέμα με τους λογαριασμούς και τη διευθέτηση των λογαριασμών στον οργανισμό. Θεωρούμε επίσης ότι είναι θετικό το συμπέρασμα της εξωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού που έγινε το 2010 από την Ernest Young. Από τα συμπεράσματα της Ernest Young, ο οργανισμός θεωρείται το αρχέτυπο ενός καλά ε, λειτουργούντος οργανισμού. Ε, υπήρχαν βέβαια κάποιες επικρίσεις ε, για το τον Οργανισμό Φαρμάκων το 2009, θεωρήσαμε ότι πρέπει να ε, δούμε κατά πόσον είναι νομότυποι και σωστοί οι λογαριασμοί, κυρίως το θέμα των ε, ε, προμηθειών για εξοπλισμό πληροφορικής. Ε, υπήρχαν μεγάλες συμβάσεις ε, πληροφορικής 30 εκατομμυρίων, 4,5 εκατομμυρίων ε, και ένας ακόμα και διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν πολύ σημαντικά σφάλματα κυρίως ως προς την αξιολόγηση τότε. Το βασικό σφάλμα ήταν μία προμήθεια 30 εκατομμυρίων ευρώ λογισμικού συστήματος, καθώς επίσης και άλλα σφάλματα, αλλά αυτό ήταν το βασικό σφάλμα το οποίο οδήγησε στο πρόβλημα. Το λάθος ήταν, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν ο οργανισμός ε, ε υπολόγισε λανθασμένα τα αποτελέσματα ενός ε, διαγωνισμού και ο οργανισμός το δέχεται ότι το ε, συνέδριο διαπίστωσε το λάθος. Ε, ο κύριος Σταυρακάκη ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια και θα πρέπει να να ζητήσουμε να εξετάζονται καλύτερε συναλλαγέ που έκανε ο οργανισμό και στην επιστολή που έστειλε ο οργανισμό ε, λένε ότι εφαρμόζουν ήδη τη σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου για να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή ε, αξιολόγηση και εμεί ε, προσβλέπουμε σε αυτού του νέου ελέγχου για του ελέγχου και του εσωτερικού λογαριασμού. Και φυσικά θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν βελτιώσει στο θέμα των προμηθειών πληροφορικής, ε, διότι κατά τα άλλα ο οργανισμός λειτουργεί πολύ καλά. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις ε, είτε δικές σας είτε των συναδέλφων σας επί του θέματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Εδώ στην αίθουσα είναι ο κύριος Πο, το εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, αλλά έχουμε και εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορούσαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και για τους δύο οργανισμούς. Και φυσικά είναι παρόν και ο κύριος Τάκαλα που εκπροσωπεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο της εργασίας, ε, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για το συντονισμό. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν σε όλες μας τις ερωτήσεις. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Κατόπιν ζήτησε να παρέμβει ε, η κυρία Μακάβεϊ. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Ο εισηγητής λοιπόν καταρχάς. Έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίζω από την πλευρά μου και το ελεγκτικό συνέδριο, τον κύριο ΣΕΑ, τους ε, διευθυντής του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων, τον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομι... ε, Αστυνομικής Ακαδημίας και το διευθυντή του... της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στον τόπο εργασίας που ε, τελικά σε αυτή τη φάση συντονίζει το δίκτυο των ε, οργανισμών. Έχω τα εξή σχόλια. Όπως σωστά αναφέρθηκε, ένα από τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα με τους οργανισμούς ήταν η μεταφορά διαφόρων κονδυλίων από χρονιά σε χρονιά. Βέβαια μπορεί να μην έχουμε μηδανική μεταφορά σαν στόχο, απ' την άλλη έχουμε όμως οργανισμούς που μεταφέρουν ποσά που ακολουθούνται από πολλά μηδενικά και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την λύση του προβλήματος. Όσον αφορά τη ΣΕΠΟΛ, την Ευρωπαϊκή Συνομική Ακαδημία, οι χθεσινές συζητήσει δυστυχώ αντί να αφορούσαν το κλείσιμο λογαριασμών της ΕΠΟΛ για το 2008, οι συζητήσει τελικά έγιναν μια συζήτηση για την απαλλαγή και τέθησαν όλα τα ζητήματα που θα ήθελα να αφήξω σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να επαναληφθεί η ίδια συζήτηση η χθεσινή, οπότε δεν θα υποβάλω ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο νέος διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας κάνει καλή δουλειά, ακολουθεί σωστό δρόμο και έκανε πολλά θετικά βήματα. Όμως, απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν ε, πολλά βήματα λοιπόν, όπως έχει και το σχέδιο δράσης, θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε εκ του σύνεγγυς της εξελίξεις. Το όσον αφορά την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κ. Σωσή αναφέρθηκε ήδη στο πρόβλημα της διαχείρισης των διαδικασιών ε, προμηθειών. Καταλαβαίνω ότι ίσως να συμβαίνουν σφάλματα, όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο οργανισμός δεν θα σε θέση να δημιουργεί σύστημα ελέγχου ούτως ώστε να αποφευχθούν ε, σφάλματα ή να, ελέγχονται, να διαπιστώνται εγκαίρως. Κυρίως αν δει κανείς ποια ποσά εμπλέκονται και τις προβληματικές διαδικασίες. Αν τα δει κανείς όλα αυτά θα δει ότι το ποσό που το προβληματικό είναι 22% του συνολικού προπολογισμού του οργανισμού. Άλλο θέμα που δημιουργεί ανησυχίες που σχετίζεται με την ενδεχόμενη ανεπαρκή χρήση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για να υπάρχει εγγύηση της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν τα προϊόντα. Ερώτημα. Η υπηρεσία έλαβε κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσει το θέμα. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σχεδιάζει μια επίσκεψη στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Διευθυντής μπορεί να μας ενημερώσει πότε. Τέλος, Εξίσου σημαντικό. Μα ανησυχούν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την ε, πρόσληψη προσωπικού που θα οδηγούσε στην πρόσληψη υποψηφίων με λιγότερα προσόντα που ίσως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα αν λάβουμε υπόψη πόσο σημαντικό ρόλο διδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κυρίως όσον αφορά το θέμα της δημόσιας υγείας. Δεύτερο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκός Οργανισμός έλαβε μέτρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έλαβε κάποια μέτρα για να καλυφθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο οργανισμούς η παραβίαση των διαδικασιών για τις δημόσιες προμήθειες είναι το βασικό πρόβλημα στην περίπτωση του ΣΥΠΟΛ, κάτι που συζητήθηκε χτες και το συζητήσαμε και στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, πρέπει να πω ότι όλοι αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο ότι βασικά ήταν χάλια κατάσταση το 2008 και μετά είδαμε ότι χάλια ήταν η κατάσταση και το 2009. Αυτό που ακούσαμε και στην αρχή των συζητήσεών μας σήμερα. Άρα έχουμε επαναλαμβανόμενες σοβαρές αδυναμίες που διαπιστώνονται. Είναι ανεξήγητο γιατί το 2009 όλες οι αδυναμίες και οι παραβιάσεις των διαδικασιών για τις δημόσιες προμήθειες συνεχίστηκαν. Όμως, θα πρέπει να εκφράσουμε ξανά τις ανησυχίες μας για τις ε, δημόσιες προμήθειες, για το πώς συνάπτονται οι συμβάσεις πώς γίνεται η πρόσληψη του προσωπικού. Και ανησυχώ λόγω ελλείψεως έρευνας μέχρι τώρα σχετικά με το γιατί οι διαδικασίες για τις ε, προμήθειες είχαν αυτές τις παραβιάσεις και δεν έγιναν έρευνες. Μας διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν έρευνες διευθυντής τη Apple, αλλά δεν έγιναν. Δεν διαπιστώθηκαν τα αίτια, δεν διαπιστώθηκαν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι το 2009 τώρα την Ευρωπαϊκή Οργανισμό Φαρμάκων, είδαμε στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου προβλήματα παραβιάσεις όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, τα κριτήρια επιλογής, τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, την Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν υπήρξε βασικά κάποια Επιτροπή Αξιολόγησης και ούτω καθεξής. Καλό το ότι και στις δύο περιπτώσεις ακούμε για προβλεπόμενες, σχεδιαζόμενες, ευκταίες τέλος πάντων βελτιώσει του 2010, όμως ας μην λησμονούμε ότι εδώ συζητούμε την απαλλαγή του 2009 και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τις ανησυχίες μας και την έλλειψη έρευνας και θα πρέπει αυτά τα κενά να εξεταστούν και οι παραβιάσεις κυρίως όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και το σχετικό σύστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος, η κυρία Γκρέτσλε και μετά η κυρία Χέρτσοκ και μετά ο κύριος Δόιτσου. Ναι, ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο. Στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες έχουμε περίπου 5.000 υπαλλήλους συνολικά προσωπικό. Α έχουμε υπόψη λοιπόν και την τάξη μεγέθου για την οποία μιλάμε. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσεύουν χρήματα από τους προπολογισμούς αυτών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, από έξι περίπου από αυτές, που έχουν περίπου πάνω από 500.000 ευρώ έσοδα τόκων το έτος. Και δεν μιλάω για το Αλικάντε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω πώς έχει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν υπάρχει αντίστοιχη διαπίστωση και για το 2009. Διότι σημαίνει, εάν αληθεύει κάτι τέτοιο, ότι τους δίνουμε πιο πολλά λεφτά από όσα χρειάζονται. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο ε, Οσίβε θα απαντήσει. Η κυρία Χέρτσοκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Είναι μεγάλη βελτίωση, πιστεύω, όσο βλέπουμε στην αστυνομική ακαδημία να λαμβάνουν χώρα, τη ΣΥΠΟΛ δηλαδή, και θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε. Πλην όμω, πρέπει να σημειώσω το εξή, ότι ενώ μιλούμε για απαλλαγή και συζητούμε το θέμα αυτό εδώ, α μην το καθιστούμε αδύνατον για του υπαλλήλου εκείνου οι οποίοι έχουν ε, την ευκαιρία ή τη βούληση να ε, πάρουν να δουλέψουν σε μια άλλη αποκεντρωμένη υπηρεσία. Μπορεί να μιλάμε για τα προβλήματα και για την αστυνομική ακαδημία κτλ. Αλλά το προσωπικό που ήταν το 2008-2009 στη ΣΥΠΟΛ έχει ίσω μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να θίξουμε. Εάν κάποιο μπορεί να πάει να κάνει μπάχαλο, λέει ο Μιλήτρια, σε μια υπηρεσία, τότε πώ μπορεί να πάει να κάνει σε μια άλλη υπηρεσία την δουλειά και εμείς να καλούμε σε λογοδοσία τους νέους ε, ε, αυτούς που ανέλαβαν μόλις καθήκοντα, τους νέους υπαλλήλου. Πώς μπορεί κάποιος δηλαδή, που ήταν πριν στην Αστυνομική Ακαδημία ε, να πάει να δουλέψει μια άλλη υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Υπάρχουν αρκετέ περιπτώσει. Και γι' αυτό το καταγγέλω. Είδαμε ανθρώπου οι οποίοι είχαν εμπλακεί τα μάλα ω υπάλληλοι τώρα να πηγαίνουν με τις ίδιες ικανότητες και γνώσεις να δουλέψουν σε άλλες υπηρεσίες. Ο κύριος Ντόιτς. Ε, Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, διακεκριμένο μέλη. Θα ήθελα να προβώ σε δύο σχόλια. Όσον αφορά την σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με την κυρία Μακοβέη και Χέρτσοκ και δεν θα επαναλάβω τα σχόλια. Συμφωνώ με τα σχόλιά τους. Έγιναν πρόσφατα τα σχόλια, μάλιστα, εδώ και 4-5 λεπτά. Το θέμα που εξετάζουμε αφορά όλους τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τους τρεις οργανισμούς που συζητούμε σήμερα και επίσης και τους άλλους οργανισμούς. Αφορά και την απαλλαγή και των άλλων οργανισμών. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι συνέβη το 2005 ή το 2010 ή τι συμβαίνει το 2011. Δεν έχει σχέση αυτό. Αυτό που θα πρέπει να ελέγξουμε είναι τι συνέβη το 2009 και αν αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, αν μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή μας ή από το Κοινοβούλιο εν γέννη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ταυτόχρονα, όσον αφορά την ΣΕΠΟΛ, η κατάσταση της ΣΕΠΟΛ δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα που ίσως μπορεί να θεωρηθεί και προηγούμενο. Αφορά το εξής. Το 2008 η οικονομική διαχείριση του οργανισμού αυτού, της Ακαδημίας αυτής, ήταν χάλια. Αυτό διαπιστώθηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο και από το Κοινοβούλιο. Και εξ αυτού απορρίψαμε την απαλλαγή, δεν χορηγήσαμε απαλλαγή. Η διαδικασία βελτιώσεων ξεκίνησε. Γνωρίζουμε τα γεγονότα. Η ίδια διαχείριση ακολουθήθηκε ουσιαστικά. Η ίδια συμπεριφορά συνεχίστηκε και το 2009. Υπάρχει όμως νέα διοίκηση από το 2010. Υπάρχει νέα διοίκηση λοιπόν στη ΣΕΠΟΛ και στόχος είναι η αλλαγή. Θέλει η νέα διοίκηση να αλλάξει τα όσα συνέβησαν το 2008 και το 2009. Είναι κατανοητό ότι συνεχώς γίνεται λόγος για την εκτέλεση του προπολογισμού προδιετίας. Αυτή όμως η χρονική κλίμακα μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε κατά πόσο ένα σφάλμα που διαπιστώθηκε προδιετίας έχει εξαλειφθεί από τη νέα διοίκηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη νέα διοίκηση της ΕΠΟΛ. Δυστυχώς όμως πρέπει να πούμε ότι και το 2009 η κατάσταση χάλια ήταν. Γνωρίζουμε όμως ότι η νέα διοίκηση ξεκίνησε κάποιες βελτιώσεις προσπάθειες βελτίωσης. Και αυτό ε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά της παρούσης διοικήσεως. Διότι και με άλλο οργανισμό μπορεί να συμβεί αυτό. Να δούμε το 2013 ότι υπήρξαν προβλήματα το 2011 Φερρυπίν αλλά ήδη θα έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες διορθώσεων των σφαλμάτων. Και μπορεί να το διαπιστώσει αυτό το κοινοβούλιο μόνο μετά από δύο χρόνια και να διαπιστώσει ότι ξεκίνησαν οι βελτιώσεις. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά λοιπόν τα φαινόμενα. Πρέπει να καθοριστούν σαφώς τα σφάλματα του 2008 και πρέπει να δούμε το πώς η νέα διοίκηση ξεκίνησε προσπάθειες, αξιόπιστες προσπάθειες για βελτιώσεις και για διόρθωση των σφαλμάτων. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σαφές όριο όσον αφορά τη ΣΕΠΟΛΑ μετά το 2010. Δεν θα αλλάχτούν βέβαια τα σφάλματα του 2008 λόγω της αλλαγής της σας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι τυχόν βελτιώσεις έχουν επέλθει. Αυτά και ευχαριστώ. Πρόεδρος, να δούμε τώρα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα υποβληθούν αρκετές ερωτήσεις προς διαφόρους, θα υπάρχουν γενικές ερωτήσεις, μετά πιο ειδικέ ερωτήσεις που θα αφορούν τη ΣΕΠΟΛ. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΟΛ είναι παρόν, ίσως όχι. Ίσως κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει κάτι για τη ΣΕΠΟΛ. Και μετά, ΕΜΕΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, και ο Α, ναι, είναι εδώ η ΣΕΠΟΛ. Συγγνώμη, τώρα σα είδα. Ναι, ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη, σα είδα τώρα. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με το ερώτημα του εισηγητή σχετικά με τα φάρμακα. Όχι. Ο κ. Τάκαλα, ο συντονιστή, ο, συντονι... Ε, που συντονίζει του άλλου οργανισμού, σα μιλήσει λοιπόν. Κ. Τάκαλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ που καλέσατε όλες τις ε, υπηρεσίες να παρούσε αυτή την τόσο σημαντική συνεδρίαση. Εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασία, αλλά ομιλώ σήμερα μόνο ω συντονιστή όλων των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Καταρχά, θα ήθελα να σημειώσω ότι έχει καθοριστική και σημασία για τι υπηρεσίε μα η καλή συνεργασία και ο συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η συμβολή στο έργο μα και ω αρχή αρμόδια και τα δημοσιονομικά ε, είναι κυριαρχεί ε, το Κοινοβούλιο για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες λαμβάνουν καθήκοντα σε διάφορους τομείς πολιτικής αρμοδιοτήτων που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει θεσπιστεί το σύνολο των υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία στην, ε, στα αποτελέσματα ανάλογα με την εντολή τους. Μπορεί να είναι διαφορετικές με οι εντολές τους και η περιγραφή τους, αλλά κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτονομία συν λογοδοσία. Κατά κύριο λόγο λοιπόν είναι υπόλογε προς το Διοικητικό του Συμβούλιο, αλλά εξίσου και στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και Μέχρι τώρα έχουν ε, στο παρελθόν εξασφαλίσει την απαλλαγή πλην μίας εξαιρέσεω όλε οι αποκεντρωμένες αρχές. Αυτό αποδεικνύει την ικανοποίηση τόσο του Συμβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου από τη δουλειά που επιτελούν αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίε, οι οποίες με πολύ μεγάλη χαρά λαμβάνουν την ενημέρωση για την απαλλαγή γιατί θεωρούν ω πολύ σημαντικές τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπαθούν να τις θέτουν σε εφαρμογή στο βέλτιστο δυνατό βαθμό όλοι μα, χρόνο το χρόνο, βήμα το βήμα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τι συστάσεις του Κοινοβουλίου. Για τα άλλα σχόλια θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο γενικά ε, σημεία προ το ελεγκτικό συνέδριο. Καταρχά για τι μεταφορέ, τα carryover. Οι υπηρεσίε γνωρίζουν ε, πολύ καλά, είναι, έχουν υπόψη του στην αρχή του ενιάφσιου χαρακτήρα του προπολογισμού και προσπαθούμε να την εφαρμόσω στο βέλτιστο δυνατό βαθμό. Όμω, πολλέ από τι δραστηριότητε μα είναι πολυετή στο χαρακτήρα, όπω και ο κύριο Σουζέ που σα εξήγησε από το ελεκτικό συνέδριο που καθόταν εδώ μπροστά μου. Συστήθηκε αυτό στην τελευταία συνεδρίαση του ελεγκτικού συνεδρίου για την απαλλαγή και με χαρά διαπιστώνω ότι και ο εισηγητή υιοθετεί την ίδια ιδέα. Δεν μπορούμε να έχουμε μηδενική δηλαδή μεταφορά κονδυλίων από τον ένα χρόνο στον άλλον. Δεν μπορεί να είναι αυτό ο στόχο μα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια συνεδρίαση, μια ε, διάσκεψη, μια ε, εκδήλωση πολιτικής προβολής λοιπά στην αρχή του χρόνου και να έχουμε ε, μόνο μέσα στον χρόνο τα κονδύλια. Πρέπει η προετοιμασία να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ή πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από ένα κονσόρσιουμ, από διάφορες ρυθμιστικές αρχές και να πάρουμε την έγκριση πριν από την τελική πληρωμή, την πληρωμή του τελικού ποσού. Άλλη εναλλακτική θα ήταν να έχουμε τις ε, μεταφορές κονδύλων, λοιπόν, το carryover. over Καλύτερος προγραμματισμός φυσικά μπορεί να αποτελέσει ένα κλειδί για τον περιορισμό του carryover, αλλά δεν μπορεί να μειώσει στο μηδέν και δεν μπορεί να αποτελέσει τη λίστα πάντα ο καλός προγραμματισμός. Όσον αφορά τώρα τους ε, ανθρώπινους μας πόρους, πρέπει να έχουμε επαρκείς ανθρώπινους πόρους ώστε να επιτελούμε το έργο μας ε, και να έχουμε πόρους για την ε, εκτέλεση των υποχρεώσεων μας έναντι του προσωπικού αυτού σε όλο το χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την αποχώρηση κάποιων μελών προσωπικού στα μισά του χρόνου ή κάποιες επιπτώσεις που έχουν αντίστοιχες, κάποια γεγονότα που έχουν αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Γι' αυτό όπως βλέπετε έχουμε υπερεκτίμηση των δαπανών του τίτλου 1. Για δε την κυρία Γκρέσλε, η οποία μάλλον έχει αποχωρήσει ήδη. Ε, αυτό που θα την ενδιαφέρει φαντάζομαι και το σχετικό με τους τόκους είναι περιορισμένης έκτασης φαινόμενο κυρίως αφορά ορισμένες ε, ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους τόκους αυτούς ούτως ή άλλως επανέρχονται στην Επιτροπή οι τόκοι. αν μείνουν τώρα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό ή αν πάνε πράγματι στο κορβανά τη Κομισιόν, αυτό είναι η αν πανε πραγματι στο γκορβανά τη Κομισιόν. Δεν μπορώ εγώ να εκφέρω γνώμη. Σημειώνω επίση ότι συμφωνούμε απολύτω ω προ την ανακύκλωση των προβλημάτων που επεσήμανε η κυρία Χέρτσοκ. Είναι κάτι το οποίο μα δυσκολεύει και είναι ένα πρόβλημα που εντοπίζονται σε αρκετέ υπηρεσίε αποκεντρωμένε, όχι μόνο στην Αστυνομική Ακαδημία. Έχει επιπλοκέ φυσικά, αλλά πρέπει να πω ότι το Φαινόμενο το εξή, δεν υπάρχει ε, είτε επίσημη δίωξη, άσκηση δίωξη, είτε επίσημη καταδίκη, δεν μπορούμε εμεί να βάλουμε κάποιον σε μαύρη λίστα μόνο και μόνο γιατί υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι στραβό. Απλώ προσπαθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, να έχουμε μια προοπτική τέλο πάντων του έχει συμβεί στο παρελθόν, που έχει πάει στραβά τι και βέβαια να κοιτάμε για το μέλλον να βελτιώσουμε τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιον σε μαύρη λίστα. Για τη λογοδοσία και το δημοσιονομικό έλεγχο. Βεβαίω θέλουμε να δασκόμαστε από την προηγούμενη εμπειρία και από τι συστάσει τη δική σα και του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο έλεγχο έχει ζωτική σημασία, δεν μπορεί όμω να υποκαταστήσει την σχέση εμπιστοσύνη ο συντονισμός των ελεκτικών ε, οργάνων και προσωπικότητων βεβαίως είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε διαχειριστικά ή διοικητικά συμβούλια, ελεγκτικό συνέδριο, εσωτερικό ε, δημοσιονομικό έλεγχο, επιτροπή αρμόδια για τον προπολογισμό, για τον ελέγχο του προπολογισμού, αρμόδιε κατ' ουσία ε, επιτροπέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τον προπολογισμό Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντίστοιχε οι συναρμόδιε γενικέ διευθύνσει, εθνικά συγγνώμη κράτη μελη Εθνικέ υπηρεσίε δηλαδή των κρατών μελών και μια σειρά άλλων ε, ε, δημοσιονομικών ελεγκτικών φορέων που κάπω θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ του. Γιατί είναι όλα στην αρμόδια. Στο ελεγκτικό συνέδριο ήδη γίνονται κάποιε προσπάθειε για περιορισμό των ελέγχων στο βαθμό όπου ο δημοσιονομικό εσωτερικό έλεγχο μια αποκεντρωμένη υπηρεσία αποδεικμένα λειτουργεί ικανοποιητικά και μπορεί τότε να προσδορίζεται κάποια προτεραιότητα και εστίαση αν πρόκειται για εξωτερικό έλεγχο που χρειάζεται. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι μια υπηρεσία λειτουργεί ικανοποιητικά μπορούμε να τη μειώσουμε τον ε, εξωτερικό έλεγχο και να την αφήσουμε στον εξωτερικό δημοσιονομικό τη έλεγχο και να επικεντρώσουμε την προσοχή μα ω προ τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο σε κάποιε άλλε υπηρεσίε που ενδεχομένω προσφέρουν περισσότερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν κοιτάμε να δούμε για καλύτερε λύσει για το μέλλον. Η αξιολόγηση η οποία ε, πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτή τη διοργανική ομάδα εργασία που έχει θεσπιστεί για τι αποκεντρωμένε υπηρεσίε επιβεβαιώνει επίση ε, την ικανοποίηση για την καλή δουλειά και τη βασική δουλειά που γίνεται σε αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Θα ήθελα και εγώ να επικεντρώσω σε αυτό και να σημειώσω τα εξή Πρώτον, συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι θα πρέπει τον έλεγχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών να τον αναπτύσσουμε κατά τρόπο οργανωμένο και συντονισμένο και με άλλου. Τα κράτη-μέλη έχουν πολύ σημαντικό ρόλο ω προ την εφαρμογή των δραστηριοτήτων των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών μέσω των διάφορων δικτύων. Δεύτερον, δεν ε, δεν κάνουν πρόσθετο έργο, δεν επαναλαμβάνουν δηλαδή έργο το οποίο ήδη πραγματοποιείται σε επίπεδο μελών, ειδικών του υπηρεσιών, υποκεντρωμένες υπηρεσίε. Έχουν ε, ανεξάρτητο και χρήσιμο έργο να προσφέρουν και θα ήθελα επίσης να επικεντρωθώ ως προς το προϊόν ε, που παράγουν οι αποκεντρωμένε υπηρεσίε, το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό και καλή ποιότητα, όσο και χρήσιμο. Πράγμα βέβαια το οποίο οφείλεται όχι μόνο στην δουλειά των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, αλλά και στην επιτυχημένη συνεργασία με άλλου φορεί, όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και οι κυβερνήσει των κρατών μελών. Επίση, παρακολουθούν οι αποκεντρωμένε ε, υπηρεσίε το έργο στη διοργανική ομάδα εργασία, στο βαθμό του δυνατού, γιατί δεν είμαστε μέλη τη ομάδα εργασία, όμω πιστεύουμε ότι μπορεί η εμπειρία μα να αποβεί χρήσιμη σε αυτήν και έτσι οπότε μπορούμε, ε, διαθέτουμε κάποιες ιδέες μέσα σε ένα έγγραφο με προτεραιότητες που μπορεί να λάβει υπόψη η ε, ομάδα εργασίας, η οργανική ομάδα εργασίας. Τα σχόλια που ακούστηκαν σήμερα βεβαίως θα τα μεταβιβάσω στο η προσεχή συνεδρίαση του, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλλον του συντονιστικού, δηλαδή τη διάσκεψη των, των διευθυντών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και θα τα λάβουμε υπόψη, βέβαια και σχέση με το Κοινοβούλιο και με το Ελεκτικό Συνέδριο. Ιδιαίτερα θα θέλω να υποχρεώσω τη σημασία που αποδίδουμε στην ε, στήριξη των θεσμικών μας εταίρων. Και πιστεύουμε ότι η λειτουργία της οργανικής ομάδας εργασίας θα συμβάλλει σε μια καλύτερη ακόμη απόδοση των εργασιών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την διεξοδικότατη παρέμβαση εξ ονόματος όλων των οργανισμών. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ε, περάσουμε στις ερωτήσεις των Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης και τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και τον εισηγητή για τα καλά του σχόλια. Πράγματι το 2009 έγινε ένα πολύ σοβαρό λάθος ε, στον οργανισμό μας ε, για τη διαδικασία προμήθειας για μια πολύ μεγάλη σύμβαση 30 εκατομμυρίων ευρώ για ένα πολυετές πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι Έχουμε μια πολύ καλά λειτουργήσα ε, υπηρεσία επαλήθευσης, έχουμε ένα εσωτερικό ελεκτή, έχουμε και μια υποπτική ε, υπηρεσία για τις συμβάσεις και τους ε, μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε να ε, διαπιστώσουμε το σφάλμα, παραβλέφθηκε και κανένας, ακόμα και οι εμπειρογνώμονές μας ε, σε θέματα πληροφορικής ε, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είχαμε ένα φύλλο Excel που θα έδινε λαθασμένα αποτελέσματα. Έγινε το λάθος, δυστυχώς δεν μπορώ να πω τίποτα για να το διορθώσω αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο νόμος του Μέρφυ χτύπησε δύο φορές. Μετά χρειάστηκε να περάσουμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις και τελικώς η σύμβαση ε, έγινε με την εταιρεία που ούτως ή άλλως θα είχε, γίνει την, ε, θα είχε κερδίσει το διαγωνισμό αν δεν είχε γίνει το λάθος ε, στο φύλλο Excel. Παρ' αυτά λοιπόν καταφέραμε να έχουμε κάποιο υλικό όφελος για τον οργανισμό. Οι επικρίσεις υπήρχαν γιατί είχαμε και λανθασμένη τεκμηρίωση και επειδή συνήθως ε, είχαμε συγκεκριμένες συμβάσεις με εταιρείε πληροφορικής. Να εξηγήσω το εξής όμως. Για τον οργανισμό μας και για τα θεσμικά όργανα, η σύναψη συμβάσεων με, για θέματα πληροφορικής ε, έχουν το εξής πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ένας οργανισμός, ένας φορέας ή οποιοδήποτε ξεκινήσει μία ε, συγκεκριμένη χρήση λογισμικού. Είτε είναι Oracle, είτε είναι Siemens, είτε Fujitsu, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας ε, ε, κλείσει μια συγκεκριμένη τεχνολογία λογισμικού, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, διότι η αλλαγή από τον έναν πάροχο στον άλλο πολύ συχνά είναι ε, τόσο δαπανηρή που είναι απαγορευτική. Πάσχουμε λοιπόν από ε, εχμαλωσία ε, σε δημόσιες προμήθειες, αν θέλετε, γι' αυτό και τόσο συχνά απλώς κάνουμε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον ίδιο πάροχο και στη συγκεκριμένη περίπτωση μας κατηγορήσαν ότι κάναμε απευθείας διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένους παρόχων υπηρεσιών. Παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε κάποια ωφέλη για, την, ε, ε, για τον οργανισμό που δεν θα είχαμε εάν είχε γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Σωστά λοιπόν ο εισηγητής είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κατά την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων μας για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για αξιολόγηση φαρμάκων, ε, το θέμα των εμπειρογνωμόνων είναι πάντα υψηλά στις προτεραιότητές μας. Έχουμε πολύ αυστηρά κριτήρια βάσει των οποίων κάνουμε ελέγχους όχι μόνο για τα μέλη του προσωπικού αλλά και ε, αποσπασμένο προσωπικό, εμπειρογνώμονας αλλά και τις οικογένειές τους πρώτου βαθμού. Σύζυγοι και παιδιά συνήθως περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία εξέτασης και ο καθής που εργάζεται ή πατάει το πόδι του στον οργανισμό φαρμάκων θα πρέπει να υπογράψει μία ε, δήλωση ε, για την ε, σύγκρουση συμφερόντων. Όσον αφορά τώρα την πρόσληψη του προσωπικού, κύριε Σιγητά, αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες βάσει του κανονισμού προσωπικού και την ε, στρέχουσας πολιτικής. Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα έχουν μηδενική αύξηση προσωπικού και μηδενική αύξηση προπολογισμού, όλα φαίνονται καλά. Αλλά υπάρχει το εξής εμείς έχουμε 170 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ δαπάνες σε φαρμακευτικά τέλη τα οποία πρέπει να δίνονται ε, κάθε μήνα και κάθε χρόνο βρισκόμαστε και με νέα νομοθεσία από τον, Ευρωπαϊκό νομοθέτη, από τον Ευρωπαίο νομοθέτη είτε είναι αυτό φαρμακοεπαγρύπνηση είτε νέα προϊόντα είτε οτιδήποτε άλλο. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό, θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε συμβασιούχους. Όπως γνωρίζετε, οι συμβασιούχοι πληρώνονται 25 με 30% λιγότερο από το υπόλοιπο προσωπικό των οργανισμών και επίσης ο κανονισμός προσωπικού των ε, ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απαιτεί να προσλαμβάνουμε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, στη χαμηλότερη δυνατή βαθμίδα για να επιτρέπεται να υπάρχει επαγγελματική εξέλιξη αλλά εμείς δεν έχουμε υπαλλήλου διαβίου στον οργανισμό. Συνήθω έχουμε πενταετή συμβάσεις, τις οποίες μπορούμε να παρατείνουμε και δυστυχώς χρειαζόμαστε ιατρικούς ή φαρμακευτικούς εμπειρογνώμονε. Κανένας εμπειρογνώμων ο οποίος έχει εμπειρία σε εργαστηριακή ανάλυση ή σε φάρμακα δεν δέχεται να έρθει στον οργανισμό ως συμβασιούχος στην κατώτερη βαθμίδα. Δεν βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσλάβουμε τους ε, εμπειρογνώμονες σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν υπάρχουν αρκετοί ιατροί, ογκολόγοι, βιοχημικοί, φαρμακοποιοί οι οποίοι είναι ναι διατεθειμένοι να έρθουν στο Λονδίνο και να εργαστούν ε, με ένα ε, με μια σύμβαση συμβασιούχου τη κατώτερη βαθμίδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας Το έχουμε ενημερώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι με τους ε, τιμέ που δίνουμε εμείς χωρί να επιβαρύνουμε περαιτέρω ε, τους ε, ευρωπαϊκούς φορείς και τους ευρωπαίους φορολογόμενους ε, θέλ, πρέπει να προσλαμβάνουμε προσωπικό σε ανώτερη βαθμίδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε θέσει ως θέμα για το μέλλον. Να σας πω και κάτι ακόμα προς τις συνέπειες. Βρισκόμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη για μας ε, θέση, πολύ καλή για το ελεγκτικό συνέδριο γιατί τη διαπίστωσε, αλλά αυτή τη δυσάρεστη ε, διαδικασία μειοδοτικών διαγωνισμών υπήρξαν συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο, έχουμε αναλάβει και τις ευθύνες μας, αλλάξαμε τη διαδικασία μειοδοτικών διαγωνισμών, συμπεριλαμβάνονται πλέον ε, στις ομάδες επιλογής και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και έχουμε αλλάξει την υπηρεσία διαχείρισης συμβάσεων και και δημοσίων προμηθειών και θεωρείται ότι είναι συνδεδευτικό φορέα σε όλε τι διαδικασίε μειοδοτικών διαγωνισμών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού, υπάρχει μια άλλη υπηρεσία που ελέγχει κάθε βήμα αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία. Όχι για να εποπτεύει το περιεχόμενο του διαγωνισμού, αλλά τη διαδικασία. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβάη νομίζω ότι είχε μία ακόμα μικρή ερώτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω στα όσα είπε η κυρία Χέρσοκ όσον αφορά εκείνους που εργάστηκαν το 2008 και 2009 στη ΣΥΠΟΛ και σε, άλλους, σε άλλες υπηρεσίες με προβλήματα και ίσως να μετακινήθηκαν και να πήγανε σε άλλες θέσεις στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα να ξέρουμε ε, έναν κατάλογο. Ποιοι πήγαν από τη ΣΥΠΟΛ σε άλλες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλους θα θέλαμε να ξέρουμε ποια ήταν η θέση τους στη δίκηση και στην εσωτερική δομή της υπηρεσίας. Ακούσαμε ότι έγινε, δεν έγινε κάποια έρευνα και δεν εντοπίστηκαν οι προσωπικές ευθύνες. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς να μετακινηθεί σε άλλους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ενώσης αν δούμε όμως τη θέση της διοίκησης, ε, καταλαβαίνουμε ποιο ποιος είναι ο ρόλος σε σχέση με τις παραβιάσεις που είδαμε. Λοιπόν, θα θέλαμε έναν κατάλογο εκείνων που μετακινήθηκαν, μετατέθηκαν και πού. Υπάρχει κάποια ερώτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να δώσετε αυτή την, αυτόν τον κατάλογο. Μπορείτε να το ελέγξετε αυτό με κάποιους άλλους. Αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο αν είχαμε αυτόν τον κατάλογο. Ο κύριος Μπόμφι λοιπόν για τη ΣΕΠΟΛ ως Μπόμφη για τη ΣΕΠΟΛ. Θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας υπευλήθησαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που είμαι ξανά εδώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να μην επαναλάβω τα όσα εξήγησα χτες. Τι κάναμε λοιπόν για να πετύχουμε την απαλλαγή του 2009 δώσαμε στον κύριο Σταυρακάκη τις κατάλληλες πληροφορίες στον εισηγητή εξηγώντας ε, κάποια μέτρα που ελήφθησαν ε, και εξηγώντα κάποια ζητήματα που τον ενδιέφεραν. Όσον αφορά τα απορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου, συμφωνούμε απόλυτα με όλα τα απορίσματα. Δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε αλλά θα κάνουμε τα δέοντα όσον αφορά τα πορίσματα. Το θέμα των προμηθειών, για να γίνει πιο κατανοητό το ζήτημα, ανακαλύφθη ότι οι προμήθειες δεν έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες. κινητή τηλεφωνία, ταξί, τα χαρτικά κλπ πριν ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την υποβολή προσφορών έπρεπε να βελτιώσω την, ε, το δυναμικό της σε πόλ, έπρεπε να ετοιμάσουμε χειρίδιο για τις προμήθειες, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό και να ξεκινήσει η διαδικασία των διαγωνισμών. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών για τα ταξί και δεν θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Δεκεμβρίου για τις επικοινωνίες της κινήτες έπρεπε να ξαναρχίσει ο διαγωνισμός, να ξανανοίξει. Είναι ο δεύτερος κύκλος όσον αφορά αυτό το διαγωνισμό. Για το προσωρινό προσωπικό και πρόσληψη από ιδιωτική εταιρεία, αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται για τα χαρτικά, για τους courier. Ε, είναι μια διαδικασία που θα θέλαμε να ολοκληρωθεί και ελπίζουμε αυτό να γίνει πριν και πριν ε, τον επόμενο έλεγχο, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς. Όσον αφορά για τις μη κανονικές προμήθειες, παράτυπες προμήθειες. Δύο άτομα, ο πρώην διευθυντής και ο γραμματέας του, ο νότερος γραμματέας του. Αυτός βγήκε στη σύνταξη, ο πρώην ε, διευθυντής δεν είναι στη θέση του πια. Αυτοί οι δύο είχαν αναμειχθεί. Και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να διεξαγάγω η αδίποτε έρευνα στην υπόθεση. Ταυτόχρονα ξεκινήσαν ιδέουσες διαδικασίες ε, έναντι των Βρετανικών αρχών και, και αυτή η διαδικασία όμως είναι εκτός των δικών μου αρμοδιοτήτων η τεκμηριωμένη γνώμη όσον αφορά, αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά τις δαπάνες σύμφωνα με, τους με το δημοσιονομικό κανονισμό για τους οικονομικούς συμβούλους κλπ. Εξέπνευσε η σύμβαση το 2009, εγώ δεν πρόσφερα παράταση των συμβάσεων. Ξεκίνησα μία εξαίρεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν μέρη συμφώνησε μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό υποχωρήσαμε όσον αφορά την πρόθεσή μας να κάνουμε μια παρέκκληση από τους δημοσιονομικούς κανόνες πέρα από το γεγονός ότι είχαμε τη νομική βάση να κάνουμε κάτι τέτοιο και βάσει της προτάσεως του Διευθυντού το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι απαιτείται συμβολή από συμβούλους και ειδικού για την εκπαίδευση όλα αυτά ε, θα καλυφθούν από τη Συμφωνία για τις Χορηγίες. Αυτή ήταν μία από τις ε, συμφωνίες που έγινε φέσος, επεξεργαστήκαμε τους κανόνες και οφείλαμε, οφείλαμε συμφωνίες πλαίσιο συνεργασίας ε, σε φορείς των κρατών μελών, τους εταίρους μας. Έχουμε 41 συμφωνίες συνεργασίας και βάσει αυτών οι περισσότερες δραστηριότητες της ΕΠΟΛ θα προσφέρονται από τις συμφωνίες για χορηγίες ε, αυτή είναι η βασική διαφορά, η βασική αλλαγή που έχει γίνει όσον αφορά τις προμήθειες. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση όσον αφορά τις συμφωνίες, τη χωρί... έχουμε τροποποιήσει τους κανονισμούς, τους δημοσιονομικούς, είναι αρμοδιότης αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά το carry over ή το carry forward των χρημάτων, τη μεταφορά πόρων των ένα χρόνο στον άλλο, Είχαμε 8,7 εκατομμύρια ευρώ το 2008, 46% μεταφέρθηκε στον επόμενο χρόνο. Το 2009 η ΣΕΠΟΛ έχει 8,6 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό και ε, πέρασε στον επόμενο χρόνο το 43% και το 2010 είχαμε 7,8 εκατομμύρια και μεταφέρουν στον επόμενο έτος φέτος 30%. Έχουμε εισαγάγει μια προσπάθεια για να διευθυνθεί η κατάσταση και εκτιμήσαμε ποιοι είναι αναγκαίοι πόροι. Μία θέλουμε να καλύψουμε τι υποχρεώσει μα όσον αφορά το πρόγραμμα στο Στοκχόλμης τη μεταφορά πόρων στον επόμενο χρόνο. Διότι η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει τη ΕΠΟΛ και θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόβλημα ανταλλαγή σύμφωνα με το πολιτικό πρόγραμμα και θέλουμε να έχουμε του πόρου. Γιατί δεν έχουμε καλύψει του πόρου, δεν έχουμε προφήσει τους πόρους ΕΠΟΛ. Πρώτα απ' όλα έγινε υπερεκτίμηση των διαφόρων εκδηλώσεων, κυρίως της εκπαιδεύσεως, της καταρτήσεως. Τα κράτη-μέλη επέμειναν η ΣΕΠΟΛ να σχεδιάζει σύμφωνα με το ότι κάθε κράτος μέσω με κουσοποιείται στην κατάρτιση. Ταυτόχρονα όμως τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι στην οικονομική θέση να στείλουν τους φοιτητές, τους μαθητέ τους σε κάθε ε, κατάρτιση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. Θεωρητικά κάθε κρατό μέλο έχει πρόσβαση στην κατάρτιση, όμως ε, οι διάφοροι εθνικοί φορεί έχουν διαφορετική οικονομική κατάσταση. Δεν έχουν τη δυνατότητα πάντα να στέλνουν ένα μέλο. Ναι, ναι, θα επιταχύνω. Ασχοληθήκαμε με όλα τα άλλα θέματα, τα ζητήματα που έθεσε το ελεκτικό συνέδριο, την υστέρηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ, εγχειρίδιο για την πρόσληψη του νέου προσωπικού, ετοιμάσαμε, φέραμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αυξήσαμε και τη διαφάνεια. Δεν είμαστε τέλειοι βέβαια ακόμα, το 2010 ήταν έτος διαχειρίσεως κρίσος και θα λήξει η κατάσταση αυτή τέλος Ιουνίου φέτος. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση όσον αφορά τις διάφορες αναπροσαρμογές. Σύμφωνα με τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου όμως πιστεύουμε ότι είμαστε όριμοι για απαλλαγή και έχουμε ανταποκριθεί σε όλες μας τις υποχρεώσεις σχετικές με την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, ο Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στον κύριο Ορσί για να ασχοληθεί με το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γκρέσλε έθεσε ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα μετρητά που έχει κάθε οργανισμός στο τέλος του έτους. Ε, αυτή είναι μια κατάσταση που διαπιστώνεται αρκετά χρόνια και την έχει διαπιστώσει το ελεκτικό συνεδρίο και προσπαθούμε να δούμε από πού έρχονται όλα αυτά τα μετρητά. Υπάρχει ε, κάποιο ισοζύγιο, γίνεται κατάλληλη διαχείριση των οικονομικών και το βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι γιατί βρίσκονται αυτά τα μετρητά ε, και κάθονται κάθε χρόνο και αν μπορεί να γίνει κάτι για τους ανθρώπους που έδωσαν αυτά τα χρήματα για τους οργανισμούς εξ αρχής. Αυτές είναι όλες οι ερωτήσεις βέβαια οι οποίες απορρέουν από την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε και η απάντηση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι θα γίνει μία ε, έρευνα, είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή για τους οργανισμούς, όπως αποχαλήφθηκε και χθε ε, στους συναδέλφους σας, και το θέμα των χρημάτων αυτών είναι ένα από αυτά τα οποία θα εξετάσουμε. Να σας πω λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το ελεγκτικό συνέδριο γνωρίζει το θέμα και θα το εξετάσει πολύ επισταμένα για όλους τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ehm, Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ούτως ή άλλως, ε, θεωρητικά η αλλως θεωρητικα έχει τελειώσει. Θα ήθελα απλώς ε, να μας δώσετε λίγα λεπτά για να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω επί του παρόντος. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σι, τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τους διευθυντές και τον συντονιστή των οργανισμών ε, για τη συνεισφορά τους και τους συναδέλφους για την ανταλλαγή απόψεων, η οποία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι εργασίε μας για σήμερα το πρωί. Θα συνεχίσουμε στις 3 ακριβώς και θα μιλήσουμε για έρευνα και ανάπτυξη σήμερα το απόγευμα. Καλή όρεξη στο επανειδή.